E Παρακαλώ καθίστε να ξεκινήσουμε την πρώτη συνεδρίασή μας ε, για το έτος 2013. Η ημερήσια διάταξη περιέχεται στον φάκελό σας και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, σχόλια, θεωρείται εγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. το γλωσσικό καθεστώς ε, καλύπτει όλες και όλους ε, τους ε, συναδέλφους. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να σας καλημερίσω. Τα μέλη, τα μέλη του Βουλής των Κοινοτήτων, του Βουλής των Λόρδων, συγγνώμη, που βρίσκονται παρόντα εδώ με κάποια αντιπροσωπεία. Να καλημερίσω φυσικά και τους υπαλλήλους της Επιτροπής μας. Θα παραμείνουν εδώ μέχρι να ξεκινήσει η συνεδρίαση αναφορικά με τον χάρτη πορείας του 2030. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω πως αύριο η συνεδρίασή μας θα ολοκληρωθεί κατά διάρκεια του πρωινού και έχει ακυρωθεί η απογευματινή. Ω εκ τούτου, οι εργασίε μα θα ξεκινήσουν σήμερα το πρωί, θα συνεχίσουν σήμερα το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν αύριο στι 12.30. Δεν θα υπάρξει απογευματινή συνεδρίαση αύριο. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω αμέσω με τον κύριο Πίπερ, που είναι εισηγητής σχετικά με τις λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους στόχους του 2020 για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τα ελαφρά οχήματα, τα καινούρια. Πόσο έχουμε, μία ώρα περίπου διάθεσή μας για συζήτηση. Δεν δίνεται απάντηση στο ερώτημα της Πρόεδρου. Κύριε Πίπερ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε, καλημέρα συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικής φύση, φυσικά και τεχνικής. Μερικές φορές αναρωτιόμαστε αν αυτέ οι τεχνικές λεπτομέρειες ε, θα πρέπει να εξεταστούν και από πολιτική σκοπιά, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο πάνω στην Ευρώπη. Πολύ συχνά υπάρχουν κάποιες προβληματικές που χρειάζεται να ε, εμβαθυθούν μέχρι την παραμικρή τους λεπτομέρεια. Και θα προσπαθήσω τώρα να δείξω τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν την Επιτροπή μας τώρα για τα νέα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Εδώ έχουμε τις ε, διατάξεις που αφορούν στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Με βάση τον κανονισμό του 2012 είχε παρουσιάσει η Κομισιόν ε, μια νομοθετική πράξη και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, πετύχαμε μια συμφωνία, δηλαδή θέλουμε να συνεργαστούμε και θα σας εξηγήσω πώς προτιθέμεθα να το πράξουμε. Υπάρχουν τέσσερις θεματικές που θα πρέπει να μας ε, εμπνεύσουν. Ε, μία φορά τα σε εκπομπές διοξιδίου του Τι γίνεται με το 2020. Ε, Εμείς θέλουμε να βάλουμε μία τάξη στις εργασίες με βάση τις υποχρεώσεις. Μετά έχουμε το ζήτημα των πιστοτικών υπερμορίων για τους υπολογισμούς σε περίπτωση που υπάρξουν καινοτόμα οχήματα τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τους απαραίτητους υπολογισμούς και δοκιμές και με βάση αυτές τις δοκιμές θα γίνουν οι υπολογισμοί στο εγγύς Και εδώ υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία. Η Κομισιόν τι προτίθεται να πράξει με αυτή την πρόταση. Καταρχήν επιβεβαιώνει τον στόχο του 142 γραμμάριων, γραμμάριων εκπομπών για τα ελαφρά οχήματα. Αυτός είναι ο στόχος που μπορούμε να επιτύχουμε το 2020. Σε περίπτωση όμως που ξεπεραστούν αυτά τα όρια, τότε ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, ποινές ε, αλλά και τις παρεκκλήσεις. Μετά το 2020 η Κομισιόν ε, θέλει ήδη από το 2014 να θέσει τους στόχους του σχετικούς προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία πριν το 2020 με στόχους πιο αυστηρούς και μετά το 2020 θα έχουμε αυτή την ε, κλιμάκωση των εργασιών και αυτές τις δεσμεύσεις. Τώρα, αυτά τα super credits πιστώσεις ε, ε, για την καινοτομία θα πρέπει να επιτευχθούν ε, μετά το 2012 με βάση το έγγραφο της Κομισιόν. Τώρα σε ό,τι φορά τις διαδικασίες δοκιμών η Κομισιόν θα φροντίσει αυτές οι διαδικασίες να συνεχιστούν. Ως εκ τούτου θα υπάρξουν νέες εξελίξεις και θα έχουμε μια νέα βάση σύμφωνα με την οποία θα ε, γίνεται ο υπολογισμός των εκπομπών. Εξετάσαμε όλες τις ε, τροπολογίες που υποβλήθηκαν και συναψίσαμε τόσο ό,τι φορά ε, τα 147 γραμμάρια και τη σχετική τροπολογία. Κατά την άποψή μας πρόκειται για ένα στόχο ιδιαίτερα φιλόδοξο. διότι προ διετία γνωρίζουμε ότι υπήρξαν ε, εκτατικές διαπραγματεύσεις και η Κομισιόν τώρα βεβαίωσε την εφικτό από τεχνική σκοπιά αυτού του στόχου. Κατ' εμάς, ο στόχος συνεχίζει να παραμένει ιδιαίτερα φιλόδοξος. Τώρα, σε ό,τι φορά αυτή την κλίμακα των εργασιών, γιατί θέλουν να την τροποποιήσουν. Δεν ισχύει, είναι πρόσφατη μάλλον η η εφαρμογή της. Εμείς ε, βλέπουμε ότι εδώ υποχρεώνουμε τη βιομηχανία να ανανεώνεται και να καινοτομεί συνεχώ. αλλά στην ουσία τη επιβάλλουν επιπλέον ε, δαπάνε. κόστο. Άρα αυτά τα ε, οχήματα θα πρέπει να βρουν και μια αγορά σε... αλλά οι πολίτες ε, θέλουν να πληρώνουν και μια σωστή, μια δίκαιη τιμή για την απόκτηση αυτών των οχημάτων. Εντάξει, είναι ένα σχεδιάγραμμα το οποίο ε, πάει καλά, ε, το μπορούσε να εφαρμοστεί. Οι στόχοι πάντως δεν είναι σίγουρα δεν είναι σίγουρο δεν είναι σαφείς Αυτά τα στοιχεία που αφορούν το 2007, άρα πριν από την ε, οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, ε, δεν αποτελούν παρά συγκυριακά στοιχεία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνάγουμε κάποια συμπεράσματα με βάση τα στοιχεία αυτά. Τώρα, να κάνω τα γραμμάρια ο στόχος, κατά θα πρέπει να παραμείνει. Τώρα, για τους στόχους με, για μετά το 2020 ακόμα δεν έχει οριμάσει το ζήτημα για να καθορίσουμε συγκεκριμένους στόχους για μετά το 2020. Έχουμε αυτά τα 147 γραμμάρια και όπως καταλαβαίνετε για τους παραγωγούς δεν είναι, για τους δεν είναι εύκολο να τροποποιούμε συνεχώς ε, τα ανώτατα όρια και να θέτουμε πιο αυστηρά διότι οι τεχνικές εξελίξεις, η νέα τεχνολογία κλπ. που έχει μπει στα σκαριά μπορεί και να μην ε, είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι χρειάζεται ένας προγραμματισμός ε, ιδιαίτερα προσεκτικός για την περίοδο μετά το 2020. Το 2018, κατά την άψή μου, θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε αναφορικά με το πώς θα λειτουργήσουμε μετά το 2020 για το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Αλλά μόνο το 2018 θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια τέτοια, ένα τέτοιο εγχείρημα. Αυτά τα super credits, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να παραμείνουν όσοι έχουν. Δεν βλέπω για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρξει αυτό το κίνητρο για τις βιομηχανίες. διότι δεν έχουν και μεγάλες επιπτώσεις στην αγορά. Άρα αυτή η διαδικασία πρέπει να διατηρηθεί. Τώρα, οι διαδικασίες ε, δοκιμών των οχημάτων. Ε, εδώ επιβάλλονται νέοι κύκλοι δοκιμών και εμεί δεν, μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτήν τη διαδικασία, διότι η Κομισιόν αυτό που θέλει να κάνει είναι να τροποποιεί και να αναθεωρεί συνεχώς ε, αυτές οι δοκιμές. αυτό δεν το επιθυμούμε, διότι νομίζουμε ότι επηρεάζει την, ε, τις βιομηχανίες, τις κατασκευαστικές αυτοκινητομηχανίες. Πάντως έχουμε ακόμα χρόνο στη διάθεσή μας ε, και θα μπορούμε να εξετάσουμε το ζήτημα περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Ναι. Γι' αυτό και σας άφησα περισσότερο χρόνο, κύριε Σιγητά, επειδή έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά είναι και πολύ εγγεγραμμένη Στο κατάλογο των αγορητών. Το λόγο έχει ο κύριος Κράμερ, σκιώδης εισηγητής ε, της Άλντε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης ε, εισηγητής ε, της ομάδα Άλντε, την Επιτροπή μα, Ο συνάδελφος Πίπερ εξέτασε πράγματι πολύ προσεκτικά το θέμα και στην ουσία συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενά του. Θα ήθελα να επαναλάβω κάπως τα λόγια του, διότι ο συμβασμός για αυτά τα ελαφρά οχήματα πραγματικά βρίσκεται στις, ε, στα σπάργανα για το στόχο 2020, δεν ξέρω θα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Παρελθόν ήμουν προδιατίας, δηλαδή ήμουν εισηγητής στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ σκληρές για να καταλήξουμε στο συμβασμό 147 γραμμαρίων. Ε, είναι σαφές ότι το 2013 αυτά τα έλαφρα οχήματα τα οποία ε, έχουν αρχίσει να ε, παράγονται τώρα βρίσκονται στην τελική φάση παραγωγής. Αν θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια ε, σταθερή πολιτική και από παραγωγή σκοπιάς θα ήταν υπεύθυνο εάν εμείς στο ζήτημα αυτό το ξαναθέσουμε για το 2020. Γνωρίζουμε ότι διεξάγονται μελέτες που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες, αλλά είναι και κάποιες άλλες μελέτες οι οποίες λένε ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. Οι, μερικές φορές οι απόψεις διήστανται. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι όλοι υπεραισιόδοξοι για τις εξελίξεις. Ε, στο έγγραφο αναφέρεται to be conform, δηλαδή να είμαστε να έχουμε συνενέσει, να, είμαστε, να έχουμε συμμορφωθεί για την εποχή, για την ε, χρονιά εκείνη. Τι να κάνουν λοιπόν για το 2020, είναι ένα θέμα που είναι κατά με ιδιαίτερα σημαντικό. Μιλάμε και για τους νέους κύκλους δοκιμών των οχημάτων. Εγώ δεν είμαι παίον ε, επί του θέματος, πρόκειται για ένα ζήτημα καθαρά μαθηματικής φύσης και όχι πολιτικής αυτός ο κύκλος των δοκιμών. Καταρχήν ο κύκλος των δοκιμών αυτός θα πρέπει να ε, εξεταστεί πριν από το να θέσουμε σε ισχύ τα, ναι, το, το τι θα λειτουργεί από το 2020 και πέρα. Εδώ πρόκειται και για μια τράπεζα δεδομένων που έχει άμεσες επιπτώσεις επί του στόχου για τον, ε, σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα όταν ε, και ο Μάρκος Πίπερ το λέει, δεν έχει ακόμα οριμάσει ο, καιρό. Πρέπει να γίνουν αυτές οι δοκιμές πριν, να αναφέρουμε ποιος θα είναι ο τελικός στόχος. Το ζήτημα είναι τεχνικής φύσης. Τώρα για τα super credits. Διότι υπάρχουν στόχοι εναλλακτικοί θα έλεγα όπως και οχήματα εναλλακτικά. Μετά το 2020, εντάξει, εγώ δεν ε, μπορώ να κάνω τον μάντι, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιο σύστημα πρόωσης ε, θα εφαρμοστεί, τι θα ισχύει. Πρέπει να έχουμε αυτές τις, αυτά τα κίνητρα για νέες, νέα είδη, νέους τύπους ε, κινητήρων. Γιατί όμως δεν γίνεται και για τα εμπορικά οχήματα μια τέτοια προσπάθεια. Αρκεί να σκεφτούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα πρέπει λοιπόν να οθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με νέα κίνητρα. Και εάν το κάνουμε για τα εμπορικά, για τα επιβατικά οχήματα θα πρέπει να γίνει και για τα φορτηγά. Πάντως νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα για την υπέρβαση των ε, θεμάτων που μας απασχολούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα ως εσκέδωση συζητής από την ECR να εκφράσω την ε, μισή μου για την εργασία που επιτέλεσε ο συνάδελφος, δεδομένου ότι έκανε μια πάρα πολύ λογική έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι τέτοιου είδου οχήματα έχουν πάρα πολύ μεγάλε και άμεσε επιπτώσει, στην ανταγωνιστικότητα και στι μικρομεσαίε καφέ ε, επιχειρήσεις. Οι οικονομικέ επιπτώσει λοιπόν μπορούν να δημιουργήσουν αβεβαιότητε ε, στον ε, βιομηχανία μα, Όχι μόνο στο επίπεδο τη αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά κυρίω όσον αφορά τι επιχειρήσει και κυρίω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε δραστηριοποιούνται πάρα πολύ στον τομέα αυτό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι 147 γραμμάρια είναι ο ανώτατος στόχος και δεν νομίζω ότι θα ήταν λογικό να ζητήσουμε περαιτέρω μείωση για τους λόγους με τους οποίους ανέφεραν οι συνάδελφοι. Όσον αφορά τους κύκλους δοκιμών θα πρέπει να συνεχιστούν διότι δεν έχουμε ακόμη αρκετά δεδομένα στη διάθεσή μας και δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις για τους οδηγούς. Τα υπερμόρια. Νομίζω ότι επίσης είναι ένα θέμα δύσκολο, διότι δεν μπορούμε ακόμη να ξέρουμε ποια θα είναι η τεχνολογία που θα έχει προτεραιότητα και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα μπορούσαν αυτά τα πιστοτικά υπερμόρια να βοηθήσουν ίσως να υπάρξει και μια κάποια σταθεροποίηση έως το 2020. Τότε θα γνωρίζουμε καλύτερα σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η τεχνολογία και ειδικά ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τα ελαφρά ΔΕΛΤΑΧ. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ λογική η προσέγγιση του συναδέλφου σε αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε την έκθεση συναδέλφου και θα να υποστηρίξουμε την ε, ε, έκθεσή του. Ευχαριστώ κύριε Τοφνόφσκι. Ο κύριος Πρόντι ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Η ε, δυστυχώ συνάδελφο Βαμπρέντ που είναι σκιώδη ε, έχει μπλοκαριστεί σε κάποιο τρένο κοντά στις Βρυξέλλες και δεν μπόρεσε να φτάσει εγκαίρως. Ως εκ τούτου με παρακάλεσε να παρέμβω στη θέση της. Ε, εν συντομία, αυτά που η συνάδελφος Βαμπραντ προτείνει είναι η υποστήριξη του στόχου για το 2025 διατηρώντας ε, τους υφιστάμενους στόχου για 2020 για των 147 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο. Φυσικά και η συνάδελφος ε, στηρίζει την αναθεώρηση του κύκλου των δοκιμών, τα test cycle, αλλά και τα super credit, τα πιστοτικά μόρια. Θεωρώ πως, ε, και αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, το αναχείρας έγγραφο αποτελεί μια πρόκληση προκειμένου να ε, παροτρύνουμε να ζητήσουμε μία πρόοδο σε ό,τι αφορά τα υβριδικά οχήματα τα οποία ήδη έχουν τεθεί στο εμπόριο. από διάφορες βιομηχανίες και θα μπορούσαν και εκεί να εφαρμοστούν τα όρια διότι σε επιτοπλίστων πρόκειται για οχήματα τα οποία κινούνται σε αστικές περιοχές και άρα θα μπορούσαν να αποφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε πρώτη. Ο κύριος Βίνταλ Κουάντρας έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι οι μεταφορές είναι, είναι υπεύθυνες για το 1 πέμπτο των ε, εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδικές το 70% αυτού του 1 πέμπτου. Η πρόταση λοιπόν της Επιτροπής είναι καλόδεχτη, διότι αναφέρεται σε ένα από τα κύρια προβλήματα και τους στόχους που θέλουμε να επιδείξουμε στα πλαίσια της πολιτικής μας στον τομέα αυτό στο 2020. Μας υπεβεβαιώνει η Επιτροπή ότι ο στόχος των 147 γραμμαρίων συγγνώμη, ανά χιλιόμετρο είναι εφικτό στα πλαίσια των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιούν και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το υποστηρίσουμε. Ο κύριο Πίπερ στην σχέδιο έκθεσή του που είναι ίσως κελισμένο να γνωρίζει ο στόχος, ότι ο στόχος αυτός για το 2020 είναι αρκετά φιλόξενος και δεν θα πρέπει να τον μεταβάλουμε η διαρκής αναθεώρηση των στόχων είναι κάτι το οποίο δημιουργεί έλλειψη εμπιστοσύνη και εξοπιστίας στη βιομηχανία. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τα μείον ώστε να είμαστε και παγκοσμίω ανταγωνιστές. Επίσης, όπως και ο κύριος Πίπερ για το 2020 συμφωνώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε την ενοποιημένη παγκόσμια διαδικασία για τα ελαφρά οχήματα, η οποία θα ολοκληρωθεί και θα θέσει τους νέους στόχους. Τελικά χαιρετίζω τα σχόλια του κυρίου Πίπερ. για το γεγονός ότι είναι σημαντικοί οι δραστηριότητες των ΜΜΕ, κυρίως στον τομέα αυτό των ελαφρών οχημάτων. και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην αυξήσουμε και τις τιμές των ε, ελαφρών φορτηγών ή άλλων των οχημάτων αυτή τη στιγμή της οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το διοξείδιο του άνθρακος για τα αυτοκίνητα είναι ένα καλό μέτρο για να μετρήσουμε πόσο οικονομικά είναι αυτά τα αυτοκίνητα. Μισό για την κλιματική αλλαγή. Ναι, όταν μιλούμε για τις εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακος, θα πρέπει να κάνουμε και διαφορετικούς υπολογισμούς και να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις εκπομπές όσο λειτουργούν τα αυτοκίνητα, αλλά και κατά την παραγωγή τους, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα διευκολύνει το σχεδιασμό για την παραγωγή τους, για την κατασκευή των αυτοκινήτων. Ένας από τους πρωτοπόρους είναι η Ιαπωνία. Δεν έχει ηγετικό ρόλο η Ευρώπη, δεδομένου ότι δεν δίνει αρκετά κίνητρα για κοινοτομίες η Ευρώπη και διότι για πολιτικούς λόγους όπως ξέρετε και η Fiat έφυγε από την Πολωνία και πήγε στην Ιταλία πάλι. Έχουμε πόρους αλλά δεν τους χρησιμοποιούμε για την καινοτομία που είναι τόσο σημαντική όσον αφορά ε, τα ελαστικά, τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων κτλ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και νέα μοντέλα που προβλέπονται για νέα αυτοκίνητα και νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να υποστηρίξει την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι κρίνω ότι είναι σωστή. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε και εσείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα άκουσα σήμερα είναι απόλυτα σωστά. Ότι δηλαδή, ιδίω ω Επιτροπή Βιομηχανία, και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, πρέπει να δώσουμε απαντήσει. Πώ θα διασφαλίσουμε δηλαδή ότι η βιομηχανία θα παραμείνει στην Ευρώπη και στο μέλλον και θα εξασφαλίζει απασχόληση. Πρέπει λοιπόν πριν από κάθε πρόσθετη επιβάρυνση να διαρωτώμεθα αν η επιβάρυνση αυτή είναι εύλογη και αν είναι το σωστό χρονικό σημείο. Μια πολιτική που κάθε χρόνο ή και κάθε εξάμεινο τροποποιεί και κάνει ακόμα πιο αυστηρά τα όρια, με την έννοια αυτή δεν είναι ευφύης. Δεν προσφέρει καμιά αξιοπιστία και δεν εξυπηρετεί τους ευρύτερους σκοπούς μας. Εμένα δεν θα μ' άρεσε να τα πούμε μεταξύ μας εδώ οι λίγοι που είμαστε, αλλά αυτή την ιδέα τελικώς να την εγγράψουμε και να την εγκρίνουμε. Να πούμε ότι θα σταματήσουμε τις διαρκείς τροποποιήσεις και επιβαρύνσεις της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρέπει να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε πλειοψηφίες ώστε αυτό το πράγμα να καταστεί σαφές και απέναντι στην Κομισιόν και απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο. Τα όσα αλέχθηκαν επί της ουσίας είναι ορθά. Πρέπει να αναμείνουμε πρώτα τις εξελίξεις και να υποστηρίξουμε τις καινοτομίες. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κανείς να καταλήξει στην ιδέα ότι οι τεχνικές αλλαγές που έχουν σαν στόχο να υποστηρίξουν, να προστατεύσουν το περιβάλλον, πώς δεν πιστώνονται σε αυτούς που τις προσφέρουν. Εδώ μιλούμε μοναχά διαρκώς για προδιαγραφές. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιατί μιλούμε ακριβώς, για τεχνικές προδιαγραφές ή για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, διότι μέχρι αποδείξεις του εναντίου κανένας δεν αμφισβητεί ότι είναι επιβλαβές το εξίο του άνθρωπος για τον άνθρωπο. Άρα αν είναι επιβλαβές, εμείς ως νομοθέτος θα πρέπει διαρκώς να προσπαθούμε να μειώσουμε τα επίπεδα ώστε να προστατεύουμε την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Συγχρόνως όμως, όντως, η βιομηχανία δεν είναι μια μηχανή την οποία μπορούμε να προσαρμόσουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και προγραμματισμός βράχει και μέσω πρόθεσμα. Μας λένε ότι θα είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό να γίνουν σημαντικές δοκιμές χωρίς να γίνει σύγκριση μεταξύ ε, αυτού του γεγονότος και το πόσο οικονομικά δαπανηρός είναι για τις κοινωνίες μας ο καρκίνος. Εάν λοιπόν δούμε αυτά τα ποσοστά και δούμε τι κοστίζει αυτό, θα δούμε ότι δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας είναι 100 φορές λιγότερες από αυτές που σημαίνει για την βιομηχανία οι πιστώσεις που παίρνουν από τις τράπεζες. Θα πρέπει λοιπόν να ψηφίζουμε κείμενα με ποσοστώσεις, με συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να κάνουμε όλο και περισσότερο ανταγωνιστική τη βιομηχανή μας σε σχέση με αυτές των υπόλοιπων κόσμων, διότι αναμφίβολα ανά τον κόσμο υπάρχει τάση τα επόμενα χρόνια να μειωθεί η ρήπανση από τις βιομηχανικές δραστηριότητες και οποιαδήποτε αρχή ε, προφύλαξης πάρουμε, βεβαίω θα είναι πλεονέκτημα σχέση με του υπολείπου. Αλλά θα πρέπει συγχρόνω να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε με παραγωγή μικροτέρων ποσότητων διοξιδίου του άνθρωπο, θα πρέπει να έχουμε ένα σφαιρικό σχέδιο. Δεν το διαθέτουμε, διότι όλο και περισσότερο φορτηγά κυκλοφορούν στους δρόμους και όπως λέει και ο συνάδελφος, είναι υπεύθυνα για τα 70% τη μόλυνση στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σφαιρικό σχέδιο που να προβλέψει συγχρόνω και τη δυνατότητα προστασία των περιλτών και ε, πιο ανταγωνιστική βιομηχανία, αλλά α μην έχουμε ψευδευτήσει θα πρέπει ε, να δούμε με μεγάλη σαφήνεια τι ακριβώς παίρνουν οι τράπεζες από τη βιομηχανία και τι κοστίζει η δημόσια υγεία για όλους μας. Ευχαριστώ κύριος Λάγκη. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Εάν θέλουμε, ειδικά για τα ελαφρά φορτηγά οχήματα, να εξετάσουμε τον κύκλο αυτό της ανανέωσης, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα 147 γραμμάρια και να τα αλλάξουμε το 2020. Αυτό νομίζω θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνενέσεως. Εδώ συμφωνώ με τον κύριο Πίπερ ότι ο στόχος που είχαμε συμφωνήσει προετών πρέπει να διατηρηθεί και να μην τον θίξουμε. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση για να υπάρξει κάποια σταθερότητα και στους κύκλους ανανέωσης των κατασκευαστών, των μοντέλων δηλαδή που παράγουν οι κατασκευαστές. Λίγες παρατηρήσεις τώρα για τα υπερμόρια και την διαδικασία και για το τι θα πρέπει ενδεχομένως να γίνει μετά το 2020. Κύριε Ρόιλ, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η πίστοση αυτή για τις ε, καινοτομίες πρέπει να θεσπιστεί έχουμε για τα επιβατηγά οχήματα. Είναι σκάνδαλο ότι έχει καταχωριστεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία και μόνη τέτοια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ δυσχερής, δυσκίνητη, πρέπει να διευκολυνθεί, να απλουστευτεί, ώστε να υπάρξουν, να προκύψουν και περισσότερες ιδέες. Και τώρα για αυτά τα super credit, κύριε Πίπερ. Εδώ πρέπει να προσφέρουμε κίνητρα για να προκληθούν περισσότερες καινοτομίες. Αυτός ο αριθμός που ακούστηκε των 100.000 οχημάτων στο σχετικά μικρό όγκο των ελαφρών φορτηγών οχημάτων, δεν ξέρω αν ο αριθμός αυτός είναι σωστός. Πρέπει να το, να επανεξετάσουμε έτσι ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένες καινοτομίες που να, έχουν, που είναι στοχευμένες. Τώρα, μετά το 2020 βεβαίω η εξέλιξη θα συνεχιστεί. Πρέπει επίσης εκεί να έχουμε σχεδιάσει συγκεκριμένα βήματα. Δεν έχει νόημα τώρα να προβλέψουμε έτσι ξεκρέμαστα έναν αριθμό, γιατί αυτό δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά κάποια καιροσκοπία. Πρέπει να καταστήσουμε σαφή την οδό μέχρι εκεί. Δηλαδή, ένα θέμα που τίθεται εδώ είναι το ερώτημα εάν θα υπάρξει νέος κύκλος δοκιμασιών συζήτηση η οποία διεξάγεται εδώ και πολύ καιρό. Πρέπει να πούμε καθαρά ότι αν μέχρι το 2015 δεν υπάρχει νέος κύκλος δοκιμασιών, τότε θα πάρουμε ως βάση τον παλαιό. Η ΔΕΜΗ κινδυνεύει αυτό να καθυστερήσει επάπειρον. Και πρέπει με τον τρόπο αυτό να δείξουμε σαφώς τον δρόμο για μετά το 2020, όπως είπα, χωρίς να κατεβάζουμε από τον αέρα κάπως ε, ξεκρέμα νούμερα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή Πίπερ, διότι η Κομισιόν θα λάβει το λόγο μετά από τη συζήτηση της προσωπικής εκθέσης. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρίως για την συμφωνία από πλευράς των συναδέλφων. Τα σημεία κριτικής που ακούστηκαν κυρίως από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και από τους πρασίνους θα προσπαθήσω να τα λάβω υπόψη για τα όσα είπε ο κ. Λάγκε, ότι ίσω ο αριθμό των 100.000 είναι κάπως υψηλό, Ασφαλώς μπορώ να το συζητήσω. Για την ίδια την διαδικασία, αν εκεί θα καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό, νομίζω ότι αυτό που προτείνω εγώ αποτελεί μια διαπραγματευτική βάση. Και αναμένω πάντως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περαιτέρω συνεργασία. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Φαίνεται πως η 30 Ιανουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι και θα έχουμε και μια συνάντηση τον Φεβρουάριο για να συζητήσουμε τροπολογίες και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται για τις 19 Μαρτίου. Και τώρα να περάσουμε στην έκθεση της κυρίας Χολ που έχει το λόγο για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στο τέλος της ε, συζήτησης των εκπομπών ε, δημιουργείται για τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρωπου ήταν ενδιαφέρον μιλήσω για οικονομικά θέματα. Υπάρχουν κοινά στοιχεία. Το σε σχέση και με τα φορτηγά. Τι πρέπει ω πιο σημαντικό στοιχείο να θυμόμαστε, ότι τα οχήματα συνεισφέρουν σε εκπομπές διοξιδίου του άθρωπου. Όλο και περισσότερο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν θέλουμε απ' την άλλη να έχουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και χρήματα θα εξοικονομήσουμε και για τους καταναλωτές και για την βιομηχανία και προστατευόμαστε και από τις εισαγωγές πετρελαίου. Η κτιμά η Επιτροπή ότι τελεία εξοικονόμηση το 2020 με 2025 θα είναι 27 δίσε και περισσότερα μέχρι το 2030 εάν μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε αυτούς τους πόρους τα αυτοκίνητα. Η πρώτη παρατήρηση λοιπόν είναι ότι καλά είναι αυτά τα νέα, διότι λειτουργεί ε, αυτός ο σχετικός ε, κανονισμός. Είναι καλύτερα και ταχύτερα τα αυτοκίνητα. Και όπως λέμε στα αγγλικά, εάν κάτι δεν χρειάζεται να το επισκευάσεις, μην το επισκευάζεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κάνουμε πολλά πράγματα έως το 2020, το οποίο για την αυτοκινητοβουλία είναι αύριο αν θέλετε, πολύ κοντά. Κάτι το οποίο προσπάθησα να κάνω είναι να δω τι θα γίνει μετά το 2020, διότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με πλαίσια των ορίζοντα του 2025 και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην προσπαθούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που προτείνει στην πρότασή της του 2020 Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τους στόχους του 2025, με απασχολεί το ότι δεν θα πρέπει να ε, συζητούμε ε, τα θέματα των δοκιμών μέχρι να έχουμε την έκθεση της UNICEF για το 2020. Ίσως ε, αυτό δεν θα το έχουμε σήμερα, αλλά το 17, το 18, αργά. Και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα, διότι το μεγάλο μήνυμα το οποίο έχουμε από την αυτοκινητοβιομηχανία είναι ότι χρειάζεται χρόνο για να προσαρμόσει τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να δούμε και να πούμε από σήμερα προς τα που θέλουμε να κατευθυνθούμε. Η αυτοκινητομία δέχεται ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε εξοικονομήσεις στον τομέα αυτό και τώρα θέλουμε να ξέρουμε ποιος θα είναι ο στόχος για το 2025. Δεν ε, θέλουμε να υπάρχουν πάρα πολλοί οι στόχοι. Υπάρχουν και άλλες αναλύσεις. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε εμείς είναι κάτι το οποίο να είναι ε, πραγματοποίησεως, δηλαδή ίσως μία μείωση κατά 20% των εκπομπών ή να έχουμε περισσότερα υβριδικά οχήματα. Το κόστος θα είναι σύμφωνα με μια τελευταία έκθεση της Ρικάρντο γύρω στα 1600 αυτοκίνητα, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι για τον όλο κύκλο ζωής του οχήματος υπάρχει ε, εξοικονόμηση πόρων για τον καταναλωτή, διότι αυτού του είδους τα οχήματα θα καταναλώνουν λιγότερη καύσιμα. Κάτι άλλο που προτείνω σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής αφορά τα υπερμόρια. Δεν θέλω να αλλάξω αυτό το οποίο λέει μέχρι το 2020 η Κομισιόν για τους λόγους που προανέφερα. Δεν νομίζω θα πρέπει να αλλάζουμε πάρα πολλά πράγματα στην πρώτη της αλλά κάτι με απασχολεί με αυτά τα πιστοτικά υπερμόρια. Η το κινητό διαμήνη χρειάζεται κίνητρα. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο να γίνουν νέα αυτοκίνητα με λιγότερες εκπομπές. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και αποδυνάμιση των στόχων. Διότι εάν ένα τέτοιο είδους αυτοκίνητο κοστίζει όσο δύο κλασικά αυτοκίνητα, αποδυναμώνεται κατά κάποιο τρόπο το στόχο. Και οι Αμερικανοί προβλέπουν κάτι τέτοιο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Με, μια πιο, με πιο ευέλικτο τρόπο. και αν μπορέσουν να επιτύχουν ε, το στόχο θα μειώσουν ε, κάπως τον τρόπο με τον οποίο παράγουν τα κλασικά αυτοκίνητα, αν το ξεπεράσουν. Αν όχι, θα πρέπει να ακολουθήσουν ένα άλλο ισχυρό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πιστοτικά υπερμόρια και μετά το 2020 θα πρέπει να έχουμε κατανοητά. Τώρα, όσον αφορά αυτό τον ε, κύκλο δοκιμών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρου των καταναλωτών για αυτό το θέμα. Και όπως σας είπα, ε, η έκθεση της UNICE δεν έχει έρθει ακόμα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναθεώρηση έγκαιρα από την Επιτροπή και να δούμε με ποιους τρόπους μπορεί αυτός ο κύκλος δοκιμών να αντικατοπτρίζει περισσότερο τους πραγματικούς, ε, τις πραγματικές συνθήκες ε, ε των αυτοκινήτων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη μελέτη και μια τελική παρατήρηση. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς μετρούμε τις εκπομπές γίνονται σύμφωνα με την μάζα. Πολύ μιλάει η Επιτροπή και για το χρήση του αποτυπώματος αντί για τη χρήση της μάζας. Διότι αν έχει Κανεί έξι παιδιά πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αυτοκίνητο. Αν παίρνει και σκι πρέπει να είναι και διαφορετικό. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι διαφορετικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Όπω σα είπα δεν πρέπει πάρα πολύ να μπερδευτούμε και να αλλάξουμε τα πράγματα στο 2020 αλλά θα πρέπει για το 2025 να δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία στην αυτοκινητοβιομηχανία για να μπορέσει να προσαρμοστεί. Ευχαριστώ. Thank you, voorzitter. Uh, mijn excuses. Er ehm, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, θα ήθελα να είμαι εδώ από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά σήμερα όπως ξέρετε είναι δύσκολα τα πράγματα στο Βέλγιο εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών. Ακούστε συνάδελφοι, εγώ πάντα έρχομαι τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Εν πάση περιπτώσει, είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα αυτό και έχει μεγάλες επιπτώσεις στην βιομηχανία. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό που διαπιστώνεται ότι θα πρέπει αυτό το βιομηχανία να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα επιχειρήματα και να τις δίνουμε τις κατάλληλες ώστε να έχουμε σωστή χρησιμοποίηση των στόχων θέλουμε να εντοπίσουμε. Και αυτό είναι σημαντικό και για μας και την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι στόχοι που έχουμε θέσει θα πρέπει να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να ξέρει ποιοι είναι οι στόχοι, είναι με από πλευράς και προ τα που κατευθυνόμεθα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει και για όλους τους ε, βιομηχάνους και είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται. Τι θέλουμε να κάνουμε εμείς, να θέσουμε στόχους για το 2020 και αργότερα και να πούμε στην αυτοκινητοβιομηχανία προς τα που θα κατευθυνθούμε. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με τους test cycle, τους κύκλους δοκιμών. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά επιστημονικά δεδομένα και αρκετές πληροφορίες για να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στην ε, τομία, στον τομέα αυτό, ώστε να ξέρουν οι πάντες περί τίνος πρόκειται. Μιλήσαμε πάρα πολύ για το eco για τον οικοσχεδιασμό και για τα πιστοτικά υπερμόρια. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους και συστήματα να τα προσαρμόζουμε στην πραγματικότητα, να χρησιμοποιούμε την ε, καινοτομία για να μην καταστρέψουμε οποιαδήποτε ε, προσπάθεια και βεβαίως να σταματήσουν οι διάφορες βιομηχανίες να παράγουν τα κλασικά αυτοκίνητα τα οποία ρηπαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε κίνητρα για την ε, αυτοκινητοβιομηχανία, να υποστηρίξουμε την καινοτομία και το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα με τον κύκλο δοκιμών με οδηγεί στο να πω ότι θα πρέπει να τον προσαρμόσουμε και αυτόν στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Merci, Madame la euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στον τύπο, σήμερα το πρωί, τον γαλλικό, αναφέρεται το κλείσιμο κάποιων εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων, όπως συνέβη με τη Ρενό, αλλά και σε άλλες πόλεις, Το θέμα που τίθεται εδώ για την Ευρώπη είναι τι είναι, τα αφήνουμε τους ε, να διαχειριστούν από μόνοι τους ε, μια κρίση ε, που προκύπτει από τον περιορισμό της ζήτησης, τον διεθνή ανταγωνισμό ή η Ευρώπη αναλαμβάνει να επιλύσει το ζήτημα συμβάλλοντας στον εξυγχρονισμό της αγοράς ε, αυτοκινήτων αλλά και στον εξυγχρονισμό της παραγωγής αυτών. Και όταν συναντάμε τους αυτοκινητοκατασκευαστές όλοι δίχως εξαίρεση μας λένε πως ε, προσοχή μην υπάρξουν νέοι κανονισμοί που θα διακυβεύουν τα συμφέροντα των βιομηχανιών μας όπως είχε συμβεί και προετών όταν ε, συζητείται ένας παρόμοιος κανονισμός. Ε, φέρουμε εδώ μια πολιτική ευθύνη. Δηλαδή δίνουμε λευκή επιταγή στους ε, αυτοκινομηχάνιους να διευθετήσουν τα προβλήματα αυτά από μόνοι τους ή τα συζητάμε για, να, για την εξέβρεση λύσης. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, είμαι υπέρ της δεύτερης επιλογής, η οποία θα βασίζεται σε όλες τις οικονομικές αναλύσεις που έγιναν και γίνονται αναφορικά με τις θετικές συνέπειες που μπορεί να έχει ε, πιο ισχυρή παρότρινση στο να κατασκευάζονται αυτοκίνητα, οχήματα τα οποία ε, εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Όταν βλέπετε τις μελέτες που έχουν γίνει ανά χώρα, διαπιστώνουμε πως η καινοτομία σε κινητήρες ψηλότερης απόδοσης και μικρότερης κατανάλωσης που εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα και καταναλώνουν λιγότερο είναι κάτι εποφελές και για τις δυνατότητες ε, καινοτομίας της αυτοκινητομηχανίας αλλά και για την απασχόληση. Είναι καλή ευκαιρία για την απασχόληση, για τη δημιουργία της θέσεων εργασίας, για το εμπορικό μας ισοζύγιο και για την εξοικονόμηση πόρων από τις εισαγωγές καυσίμων. Αυτή είναι λοιπόν η καλύτερη λύση, εκτός φυσικά αν προσανατολιστούμε προς την εξαγωγή μοντέλων που αφορούν ε, πελατεία υψηλή Λοιπόν, εμείς ε, είμαστε υπέρ της αναθεώρησης του στόχου του 2020 για τα 80 γραμμάρια. Θα το ονομάζουμε ευελιξία, αλλά κανονικά πρόκειται για καταργήσεις ε, Φυσικά στηρίζουμε την αναθεώρηση των ε, δοκιμών που γίνονται για τις εκπομπές, διότι δυστυχώς όλα αυτά ε, οδηγούν στο να διατηρήσουμε το status quo παρά να υπάρχει ανανέωση και γίνοντα με ευχαριστώ και τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στο προηγούμενο θέμα της της διάταξης συζητήσαμε ένα παρόμοιο σύνολο ας πούμε ιδεών. Τώρα είναι λίγο διαφορετικό. Και βέβαια είναι δύσκολη η προσπάθεια να καταλήξουμε στη σωστή απόφαση. Πρέπει να είμαστε άραγε πιο φιλόδοξοι στην επίσημη ας πούμε πλευρά, δηλαδή με την έννοια της επιβολής μέτρων ή πρέπει να παραχωρήσουμε περισσότερο χώρο, περισσότερη ελευθερία στην αγορά. Να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ο κόσμος θέλει να αγοράσει οικονομικά αυτοκίνητα. Όλοι αντιμετωπίζουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης. Η συζήτηση στρέφεται γύρω από το τι είναι καλύτερα τελικά ως τακτικός ελιγμός. Η δική μου σύσταση είναι προσοχή. Να μην υπερβάλλουμε με τα διοικητικά μέτρα. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι δεν πρέπει να στατώνουμε τους στόχους που έχουμε επιβάλει για το 2020, βάζοντας έτσι ένα στοιχείο ανασφάλειας ε, για την αυτοκινητοβιομηχανία, γιατί η παραγωγοί, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν είναι μόνο αυτοί που ενδεχομένω θίγονται, γιατί υπάρχουν και όλοι οι προμηθευτές, υπεργολάβοι, αλλά επίσης οι αυτοκινητοβιομηχανίε ε, ασχολούνται και με άλλου είδους παραγωγές. Γι' αυτό συστήνω προσοχή και αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά την θέσπιση στόχων για μετά το 2020 να παρακολουθήσουμε προσεκτικά τις εξελίξεις. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων καμιά φορά αναγκάζονται να κλείσουν. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζουν μόνο τις οικονομικές πιέσεις που όλοι βλέπουμε λόγω της κρίσης στην Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, καμιά φορά αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν και τις ανάγκες που επιβάλλουν οι κύκλοι ανανέωσης των μοντέλων τους. Πρέπει να δώσουμε περιθώριο στους κατασκευαστές να αναζητήσουν νέες τεχνολογίες. Αυτά τα κίνητρα πρέπει να διατηρηθούν. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε διοικητικά, ας πούμε, άνωθεν ότι θα, θα, κατασκευαστούν περισσότερα υβριδικά ή ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κτλ. Ίσως να προκύψει μια νέα τεχνολογία που να επιτρέψει όλους να κινηθούν ταχύτερα προς τα εμπρός. Ας μην λοιπόν τους επιβάλλουμε τι να κάνουν. Η δική μου πολιτική ομάδα πάντοτε προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ του να είμαστε μεν φιλόδοξοι, όχι όμως με τρόπο που να οδηγεί σε δυσκολίες την αυτοκινητοβιομηχανία. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς να τους κινητοποιήσουμε, τους κατασκευαστές, να παρακολουθούμε, να παρατηρούμε τις εξελίξεις τα όρια δε των εκπομπών που έχουν θεσπιστεί πρέπει να επικυρωθούν, να επιβεβαιωθούν, να αποφύγουμε οποιασδήποτε δραματικές αλλαγές που επιβαρύνουν την αυτοκίνητο βιομηχανία. Ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα και, και τους πρασίνους που λένε «Ω, ρυθμίσεις επιρυθμίσεων όλο και ψηλότεροι και αυστηρότεροι στόχοι κλπ. Αν συνεχίσουμε να επιβάλλουμε όμως αυτά στην Ευρώπη και δεν μας ακολουθεί κανείς, τότε και οι αγορές θα αντιδράσουν. Και η συνολική παγκόσμια παραγωγή, η θέση μάλλον της παραγωγής μας παγκόσμια θα αποδυναμωθεί. Έτσι λοιπόν, αυτά που προτείνουν οι πράσινοι και εν μέρη και οι σοσιαλδημοκράτες δεν βοηθούν πολύ. η συνάδελφό μα που μίλησε πριν εκπροσωπεί τον κύριο Μπρεζίνα, ο οποίο έχει συντάξει, είναι απόν σήμερα. Υπάρχει λοιπόν μια πρώτη προσωπική παρατήρηση. Κυρία Χόλμ, για την κυρία Χόλμ αναφέρομαι τώρα. Ευχαριστώ πολύ που μα υποστηρίζετε για τα 95 γραμμάρια μέχρι το 2020. Μετά όμω η πρότασή σα και τώρα παραθέτω αυτό που λέει ο κ. Μπριζίνα, δηλαδή να φτάσουμε μέχρι το 2025 στα 70 γραμμάρια, αυτό είναι υπερβολικά πρόημο. Όταν ανησυχείτε εσείς για τις οικογένειες με τα μεγάλα αυτοκίνητα, τότε πραγματικά αναβλύζουν δάκρυα στα μάτια μου, αλλά και θέλετε μετά να βάλετε και τα σκι. Εγώ ανησυχώ περισσότερο για οι οικογένειες ε, με παιδιά που δεν έχουν τα μέσα καν να αγοράσουν ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Και ω ε, σχετικά ε, οι οικογένειε με περιορισμένη, α πούμε, με περιορισμένο εισόδημα, πρέπει και, αυτοί να έχουν, και αυτές να έχουν το, τη δυνατότητα να προμηθευτούν ένα αυτοκίνητο που να του εξυπηρετεί. Εμεί δεν είμαστε λοιπόν σύμφωνοι από τώρα να θεσπιστεί ο στόχο των 70 γραμμαρίων μέχρι το 2025. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερε πληροφορίε και το πολύ ίσως το 2015 μπορεί να διατυπωθεί τέτοιο στόχο. Ωστόσο μέχρι τότε πρέπει να αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ε, παγκόσμιας εναρμονισμένης ε, δοκιμασίας για τα ελαφρά οχήματα. Τώρα, για τα ε, super credits αποτελούν και αυτά κίνητρο για την βιομηχανία και εμείς θέλουμε να διατηρηθούν και μετά το 2020. Οι περιορισμοί που προτείνεται κυρία Χόλμ στην έκθεση είναι, πώς να πω, δεν μας βοηθούν. Δεν μας βοηθούν. Θα πρέπει να θα, να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβασμού στην περαιτέρω πορεία. Ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Κύριε Λάγκε. Ευχαριστώ. Κύριε Πίπερ, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το διοξίδιο του άνθρακα έχει στην ουσία ενισχύσει την θέση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Βλέπουμε ότι και άλλοι παγκοσμίω ακολουθούν, αλλά και βλέπουμε και τα μερίδια τη Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία τη διεθνή πωλήση αυτοκινήτων και δεν μπορεί κανεί να παραπονείται σχετικά. Τώρα, για του στόχου. Πάλι εδώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι πρέπει να περιμένουμε αυτόν τον περίφημο παγκόσμιο κύκλο δοκιμασιών. Αυτά τα πράγματα έχουν πολύ σχέση και με τον ανταγωνισμό. Αν θα συμφωνήσουν δηλαδή οι Αμερικανοί σε ένα παγκόσμιο τέτοιο σύστημα ή όχι για να προαχθεί η προοπτική και μετά το 2020, το 2015 σταματάει η συζήτηση για τον παγκόσμιο κύκλο δοκιμασιών και μένουμε στον παλαιό κύκλο. Γιατί αλλιώ ε, αναβάλλεται, καθυστερεί η υπόθεση αυτή επάπειρον. Και για τα φορτηγά αυτοκίνητα και για τις μοτοσυκλέτες είχαμε κάνει τη συζήτηση αυτή για τον παγκόσμιο κύκλο. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι και εδώ η διαδικασία για το πώς θα προχωρήσουμε μετά το 2020 πρέπει να ξεκαθαριστεί από τώρα. Έχουμε μια προοπτική μέχρι το 2050 στην Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές προς τα που θέλουμε να κατευθυνθούμε δηλαδή και στο μεταξύ πρέπει να ρυθμίσουμε τα μέχρι τότε βήματα. Τώρα για τα super credit. Κύριε Πίπερ και εδώ δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να τα συνδέσουμε με τον όγκο παραγωγής διότι ε, έχουμε και διαφόρους κατασκευαστές. Ένας μικρός κατασκευαστής που παράγει περιορισμένο αριθμό οχημάτων θα τα αντιμετωπίσει ευκολότερα από ένα μεγάλο κατασκευαστή. Ίσως είναι καλύτερα να συνδεθεί με την αξία των πωλήσεων. Και για την eco-innovation πρέπει εδώ η διαδικασία ασφαλώς να απλουστευτεί έτσι ώστε οι καινοτομίες αυτές να περνούν στην αγορά ταχύτερα. Έθεσα κάποιες ερωτήσεις στην Κομισιόν γύρω από το ερώτημα για ποιο λόγο τα τελευταία χρόνια εγκρίθηκε μια μόνο τέτοια. Ε, η Κομισιόν υποσχεθεί ότι θα εγκύψει στο θέμα. Αλλιώς πρέπει να το επανεξετάσουμε και να το περιλάβουμε στην νομοθεσία. Άρα, ξεκάθαροι κανόνες για τα super credit, καθώς επίσης ξεκάθαροι κανόνες για τα βήματα που πρέπει να γίνουν μετά από το 2020. Ο Ελάτε μαζί μου ξανά στο 2008. Τότε εγώ ήμουν εισηγητή για τον πρώτο συμβιβασμό με τον στόχο των 95 γραμμαρίων. Είχαμε πει τότε ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξο ο στόχο ότι θα φέρει μεγάλε αναστατώσει. καταφέραμε και τα περάσαμε τότε ως χριστιανοδημοκράτες και όπως είπε και ο κύριος Λάγκη, ο οποίος δεν ήταν παρόν εδώ τότε ως Ευρωβουλευτής, αλλά το επιβεβαιώνει τώρα, αποδείχθηκε ότι έκανε καλό στην ανταγωνιστικότητα. Τώρα έχω πέντε σχόλια. Πρώτα, η πιο αυστηρή θέσπιση στόχων έχει σχέση με τη βιομηχανική πολιτική για άλλα τα προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα, τα οποία από τις διεθνείς μεταφορές μέχρι τις εναέρειες μεταφορές μέχρι τώρα δεν έχουν επιτύχει, δεν έχει εμφανιστεί καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα, οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις ε, αποδείχθηκαν επιτυχημένες ήταν λόγω του ότι έγινε συνδυασμός τεχνολογικών κινήτρων, eco-innovation και ούτω καθεξής με μακροπρόθεσμους στόχους. Εάν τώρα, και αυτό είναι το ερώτημα, αν θέλουμε τώρα νέο μακροπρόθεσμο στόχο πέντε χρόνια μετά από το πολύ φιλόδοξο στόχο των 95 γραμμαρίων, όπως προτείνει τώρα η Κομισιόν και η κυρία Χόλμ τα κάνει ακόμα πιο αυστηρά, τότε βάζουμε δυσκολίες όχι μόνο στη βιομηχανία, αλλά εμφανιζόμαστε σαν δήθεν να μπορούμε καλύτερα και από τους μηχανικούς να αποφασίσουμε ποια, είναι τεχνικά, ποια πράγματα είναι τεχνικά εφικτά. Γιατί 70 γραμμάρια μέχρι το 2025 σημαίνει ότι κανένα φορτηγό που θα παράγεται μέχρι τότε δεν θα μπορεί να καταναλώνει πάνω από 3 λίτρα καυσίμου ανά 100 χιλιόμετρα. Αυτό είναι ψευδέστηση. Είναι αδύνατο να το επιτύχει η ε, ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Και όλες αυτοί, όλοι αυτοί οι θρήνοι που ακούγονται εδώ για τα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, για τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή, δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθούν εάν βάλουμε τέτοιους υπερβολικούς στόχους. Τώρα για την κυρία Ρολ, η οποία ήδη το 2008 συγγνώμη, έλεγε αυτά για το ίχνος ήδη τότε προτείνονταν 75 γραμμάρια για τον κύκλο δοκιμασιών, για τις ε, καμπύλες και ούτε καθεξής. Είχαμε καταλήξει τότε σε ένα συμβασμό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος απολύτως εν ώψη των μεγάλων επιτυχιών της αυτοκινητοβιομηχανίας με την υφιστάμενη οδηγία να τα κάνουμε ακόμα πιο αυστηρά και δεν καταλαβαίνω και την Κομισιόν. Αφενός η Κομισιόν ζητεί μια συνεπή βιομηχανική πολιτική, από την άλλη μεριά άλλα χαρτοφυλάκια της Κομισιόν κάνουν τα αντίθετα. Αφενός κλαίνε για την απώλεια τη βιομηχανία από την Ευρώπη, την αποχώρηση από την Ευρώπη και από την άλλη μεριά κάνουν ό,τι μπορούν να δυσκολέψουν. Γι' αυτό θα συμφωνήσω με τους Πίπερ, Πριτσίντα, Λάγκε και άλλους που είπαν ότι πρέπει να φανούμε με τριοπαθείς και αν διατυπώσουμε μακροπρόθεσμο στόχο δεν μπορεί αυτός να είναι 5 χρόνια μετά να πω τον υφιστάμενο στόχο. Ας πούμε 15 χρόνια ή τέλο πάντων ας δείξουμε φαντασία. Ας πούμε 70, 70 γραμμάρια το 2035, όχι 70 το 2020. Ο Κουαράς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση της Κομισιόν για την τροποποίηση του κανονισμού προκειμένου να διορίζουν ε, διαδικασίες για τη μείωση των εκπομπών είναι παρόμοια με την προηγούμενο έκθεση που εξετάσαμε και υπάρχουν ως εκ τούτου πολλά στοιχεία κοινά και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα στις συζητήσεις μας για το έργο μας, θα πρότεινα, εάν φυσικά οι συντονιστές και οι σκιώδεις συμφωνούν, ότι στο μέλλον για, αυτά, για αυτούς τους δύο κανονισμούς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κοινή συζήτηση. Γιατί πάνω κάτω πρόκειται περί του αυτού θέματος. Θα μπορούσαμε να το θέσουμε λοιπόν στο αυτό σημείο στην μεσαδιάταξη. Φυσικά αυτή είναι μια πρόταση που θέλω να κάνω. Τώρα, σχετικά με την ε, γνώμη της κυρίας Χόλς, τη γνωμοδότηση μάλλον, αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ότι η Κομισιόν θα πρέπει με τα κρατημέρια τη της περιφέρειας να δημιουργήσει κίνητρα για οχήματα ιδιαίτερα χαμηλών ε, εκπομπών. Ευχαριστήρια θα πρέπει να δώσουμε στην Φιώνα Χολ που μας ε, προειδοποιεί για τις διαφορές που υπάρχουν σχετικά με την καταγραφή των εκπομπών. Διότι παρεμποδίζει την σωστή εκτίμηση του προβλήματος. Αλλά κατά την άποψή μου θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των δοκιμών που γίνονται δεν θα ήταν ε, λογικό να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα τώρα και ένα άλλο για αυτό που προτείνει η Κομισιόν για το 2015 και ένα άλλο για ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα όταν αυτό θα είναι έτοιμο. Δεν πρέπει λοιπόν να βιαστούμε. και δεν βλέπω το λόγο να θέσουμε στόχο για το 2025 σε αυτή την πρόταση. Τώρα μιλάμε για τους στόχους του 2020. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε στόχους για το 2025 σε αυτό το φάση. Οι βιομηχανίες γνωρίζουν την κατεύθυνση που ακολουθούμε και μια που έχουμε έναν φιλόδοξο στόχο θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην επίτευξη αυτού του στόχου και να αφήσουμε τη συζήτηση για τους νέους στόχους όταν θα έχουμε καλύτερη γνώση περί του υπολογισμού των εκπομπών. Αυτά τα δύο πράγματα είχα να πω, Φιώνα. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστώ την Φιώνα Χολ για τη γνωμοδότηση. Συζητούμε για το τι θα γίνει μετά το 2020. Χαίρομαι που στη γνωμοδότησή της επιβεβαιώνει τα 95 γραμμάρια. Εδώ υπάρχει ένα επιχείρημα ωστόσο, το οποίο πλανάται ως φάντασμα και εδώ στην αίθουσά μας αλλά και στην έκθεση. Δεν υπάρχει αυτόματη διασύνδεση μεταξύ φιλόδοξων στόχων ε, στη, για την προσέγγιση του περιβάλλοντος και την επιτυχία των αυτοκινητοβιομηχανιών. Ο Ευρωπαίος τσάμπιον της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι αυτός που έχει και τα μεγαλύτερα υπαρξιακά προβλήματα. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια για την επιτυχία κάποιων αυτοκινήτων μεταξύ των καταναλωτών. Και αν βάλουμε διάφορε νομοθεσίε τη μια δίπλα στην άλλη, που είναι δύσκολο να συγκριθούν, αν όμω όμως προσαρμοστούν, α πούμε, τότε θα δούμε ότι η Ευρώπη είναι ο πρωταθλητή στην καταπολέμηση τη εκπομπή των διοξιδίων του άνθρακα. Όταν σήμερα μιλούμε για στόχους για μετά το 2020, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και κάποια όρια της φυσικής για το τι είναι δυνατόν να γίνει το ότι είναι εφικτό. Έχουμε σήμερα σχεδόν 100% κινητήρες εσωτερικής καύσεως στην αγορά. Με την τεχνολογία που διαδέτουμε σήμερα και που είναι δυνατόν να την πληρώσει ο καταναλωτής και είναι και διατεθειμένος να την πληρώσει, τέτοιοι στόχοι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Τώρα, πού θα βρεθεί η νέα τεχνολογία. Αυτά πρέπει να γίνουν αντικείμενο νέων ερευνών. Τώρα, πού θα φτάσει το όριο, μπορεί να φτάσει στα 75, στα 70, στα 60 γραμμάρια. Αλλά δεν μπορεί να το αποφασίσει αυτό η Επιτροπή Βιομηχανίας. Ας συζητήσετε και εσείς και με την κυρία Βαν Μπρέμπτ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτό το ερώτημα στη βάση ποιο κύκλο δοκιμασιών θα θεσπίσουμε όρια μετά το 2020. Εάν υπάρξει νέος κύκλος δοκιμασιών, τότε βέβαια πρέπει να ληφθεί ως βάση. Αν όμως δεν υπάρξει, τότε πρέπει να λάβουμε τον παλαιό ως βάση. Δεν μπορούμε όμως να θεσπίσουμε νέους στόχους χωρίς να γνωρίζουμε στη βάση ποιων κύκλων δοκιμασιών. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι μαθηματικά, διασυνδέονται. Δεν είναι πολιτική απόφαση. Πρέπει να είναι πρώτα ξεκάθαρο αυτό για να υπάρχει άλλωστε και κάποια σαφήνεια απέναντι στην βιομηχανία. η Κομισιόν για τα δύο κείμενα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους κύριους Πίπερ και Χολ για τις, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων. Ας αρχίσουμε με τη γνωμοδότηση για τα φορτηγά, τα μικρά φορτηγά. Σχόλια για δύο πράγματα. Πρώτα για την διαδικασία επανεξέτασης και ύστερα για τα υπερμόρια, τα super credit. Σε ό,τι αφορά την επανεξέταση, η Κομισιόν είπε ότι θα υποβάλει το 2014 σχέδιο διαδικασίας για μακροπρόθεσμο στόχους μετά το 2020. Όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Διότι ο στόχος του 2020 για τα 147 γραμμάρια είχε γίνει προ 8 ετών και είχαμε δώσει για τα, είχαμε προσφέρει 9 χρόνια στους κατασκευαστές γνωρίζοντας ότι η κύκλη ανανέωση των μοντέλων είναι μεγαλύτερη από ό,τι για τα επιβατικά οχήματα, το ίδιο πάμε να κάνουμε και τώρα. Για τα επόμενα 10 χρόνια, δίνοντα του ε, κατασκευαστέ και μια ασφάλεια. Αυτό είναι σημαντικό. Επειδή άλλωστε έχουμε και παγκόσμια βιομηχανία η οποία ε, ανταγωνίζεται, οι διάφοροι και στην παγκόσμια αγορά. Ακούσαμε επίση διαφόρου ευρωβουλευτέ να μιλούν για τον οδικό χάρτη και τη λευκή βίβλο. Ναι, είναι πράγματι ότι, είναι πράγματι αληθές ότι είναι φιλόδοξοι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Έχουμε ωστόσο μια ε, συνολική μακροπρόθεσμη πρόπτικη και σωστό είναι αυτό για να γνωρίζει η βιομηχανία προς τα που κατευθυνόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πάμε να θεσπίσουμε τους μελλοντικού μακροπρόθεσμους στόχους. Τώρα, για τα super credit. Ας υπενθυμίσω ότι για το 2017 έχουμε 117 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο. Και αυτό που έχουμε σήμερα είναι το impact assessment. Για το 2010 είχαμε φτάσει στα 180 γραμμάρια. Άρα μεγάλη απόσταση. Τώρα, εμείς βλέπουμε στην ουσία να αποδυναμώνεται ο στόχος αυτός σε διαφόρους τομείς. Αφενός βλέπουμε μια αποδυνάμωση, διότι το κατόφλι φεύγει από τα 50 γραμμάρια και πάει σε ένα μέσον όρο 87 γραμμαρίων. Δεύτερο, διότι έχουμε βάλει ένα πολλαπλασιαστή για το 2017. Τρίτο, γιατί γιατί έχουμε συμφωνήσει άλλωστε προ δύο ετών από τα 25.000 οχήματα στα 100.000 οχήματα. Περίπου δηλαδή στο επίπεδο πωλήσεων της Volkswagen ή της Daimler-Benz. Άρα μειώνουμε τον στόχο αυτό στην πραγματικότητα, που δυναμώνουμε τον στόχο αυτό στην πραγματικότητα με τρόπο που γίνεται υλοποιήσιμος κατά τη γνώμη μας. Τώρα, για τους μακροπρόθεσμους στόχους μετά το 2020, εμείς θεωρούμε ότι είναι δυνατόν αυτό με ένα πρόσθετο κόστος 450 ευρώ ανά ε, φορτηγό, ανά φορτηγάκι τέλος πάντων, βαν. Αυτό σημαίνει ότι θα εκπέμπονται μεταξύ 2020 και 2030 2 εκατομμύρια τόνοι ε, καυσαερίων παραπάνω. Επίσης σημαντικό είναι να θυμηθούμε και τι λέει European Small Business Alliance, Carlis κλπ που είπαν δηλαδή σε διάφορα μέλη της Επιτροπής σας και που ζητούν οι φορείς αυτοί πιο φιλόδοξους στόχους. 118 γραμμαρίων γιατί αυτό θα τους ε, επιτρέψει να κάνουν εξοικονομήσεις. Η ίδια η βιομηχανία λοιπόν ζητεί να γίνει πιο σφιχτή η στόχη. Δεύτερο, έρχομαι σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και για τις δύο γνωμοδοτήσεις και για τα αυτοκίνητα και για τα ελαφρά φορτηγά. Το test cycle, ο κύκλος δοκιμασιών που έχουμε τώρα, τον ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμασιών, τον οποίο γνωρίζουν και τον έχουν συνηθίσει οι κατασκευαστές και πάση περιπτώσει αυτόν έχουμε σήμερα. Για πολλά χρόνια το WLTP έχει αναπτυχθεί υπό την αιγίδα των Ενωμένων Εθνών και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ φέτος θα δοθεί τελική μορφή στη διαδικασία UNICE και του χρόνου ή το 2015 θα γίνουν και οι νομοθετικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε λοιπόν μια περίοδο χρόνου μετά όπου αυτό θα μπει σε πλήρη εφαρμογή. Και είπαμε και για τις δύο προτάσεις ότι θα προσαρμόσουμε τον κύκλο δοκιμασιών για να είναι το ίδιο αυστηρός και δεν θα προχωρήσουμε περισσότερο πρέπει να γνωρίζουμε καλώς, να, μην, αποφύγουμε να γίνει ε, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε αντιπερισπασμός από τη UNICE ή WLTP. Τώρα, για τους μακροπρόθεσμους στόχους. Είναι σαφές ότι οι Ενωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ένα στόχο για το 2025. Επίσης, τα 70 γραμμάρια για το 2025 είναι φιλόδοξο, είναι 6% μείωση ανά έτος είναι όμως δυνατό και με την υβριδοποίηση η οποία θα προχωρήσει από πλευράς πολλών κατασκευαστών. Το impact assessment της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη εξετάσει τα 70 γραμμάρια το 2020 ασφαλώς και προκύπτει ένα κόστος για τους κατασκευαστές αλλά νομίζουμε ότι για ένα μεσαίο αυτοκίνητο το συνολικό κόστος ε, θα ε, εξισορροπηθεί από το συνολικό όφελος. Για τα super credit τώρα, για τα αυτοκίνητα είναι σωστό ότι η Κομισιόν, η Κομισιόν είναι σαφές από την ε, ε, μελέτη επιπτώσεων που έκανε, αγωνίστηκε για τα super credit. Βλέπουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα, είναι ουδέτερο ό,τι αφορά την τεχνολογία, προσφέρει ένα κίνητρο στους ε, κατασκευαστές για να αυξήσουν τις πωλήσει τους και θα αυξηθούν και εξοικονομήσεις από το 2020 μέχρι το 2030. Ωστόσο, Εάν υπάρξουν ε, υψηλότεροι πολλαπλασιαστέ από αυτού που προτείνει η Κομισιόν, τότε το αποτέλεσμα στι εξοικονομήσει θα είναι χαμηλότερο. Τώρα για το ίχνος, footprint, το εξετάσαμε προσεκτικά στην μελέτη επιπτώσεων. Αναγνωρίζουμε τη σχέση κόστους-οφέλους. Ωστόσο, να δοθεί η επιλογή στους κατασκευαστές από τώρα μέχρι το 2020 θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ε, υπό ορισμένε ε, οπτικές γωνιές για για την περίοδο μετά το 2020 είπαμε και στους stakeholder και στη βιομηχανία ότι αυτό πρέπει να επαναξεταστεί διότι πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα πλήρως τα θετικά και αρνητικά του στοιχεία. Τέλος για τις eco-innovation είναι σωστό ότι η εργασία συνεχίζεται Όντως υπήρξε μία εγκεκριμένη eco-innovation, όμως άλλες βρίσκονται αυτή τη στιγμή που επεξεργασία και θα έχουμε ε, σύντομα εξελίξεις να σας πούμε. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά δυστυχώς ε, με... έχουμε καθαρίσει και σε αυτό, έχουμε, ξε... έχουμε καθυστερήσει, συγγνώμη και πρέπει να βιαστούμε. Δώσω τον λόγο στην συνάδελφο Όλου και μετά θα συνεχίσουμε εμείς τη διάταξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους που με βοήθησαν πολύ. Χαίρομαι διότι πιστεύω ότι υπάρχει συνένεση ότι δεν θα πρέπει με τους ε, στόχους και τη βασική δομή του 2020 να αλλάξουν πολλά πράγματα. Χαίρομαι που συμφωνήσετε. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν του συναδέλφου. Το θέμα της παγκόσμια ανταγωνιστικότητας. Συμφωνώ με τον κύριο Λάγκε. Θα πρέπει πραγματικά να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να μην μείνουμε πίσω. Διότι αυτό δεν είναι κάτι που κάνει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό που δεν θέλουμε είναι η δική μας βιομηχανία να καθυστερήσει και να μην είναι αντιγωνιστική στις αγορές οι οποίες όλο και περισσότερο για θέματα εκπομπών ε, ε, διοξιδίου του άνθρακος είναι πιο αυστηρές. Τώρα, η Επιτροπή τώρα μόλις επιβεβαίωσε ότι το κόστος αγοράς μπορεί να είναι υψηλότερο, αλλά για τον κύκλο, σε όλο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου κάνετε οικονομίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από τη βιομηχανία και για τους κατανοτές, διότι γιατί παραπονούνται συνέχεια κάθε μέρα. Πόσο ακριβά κοστίζει αυτή τη στιγμή ε, η βενζίνη ή το ε, πετρέλαιο. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να με απασχολεί, διότι πρόκειται για χρήματα τα οποία χάνονται για όλες τις οικονομίες. Αν δείτε λοιπόν τι κάνετε, ε, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε και τους καταναλωτές να βοηθάτε για διάρκεια όλου του κύκλου ζωής του αυτοκινήτου και τη βιομηχανία. Είπε ο κ. Λάγκη ότι για να, θα πρέπει να κάνουμε κάτι σαφές. Σήμερα μιλούμε για ένα στόχο, ο οποίος είναι ο μέσος όρος δεν είπα ότι όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν φτάσει έως το 2025 σε εκπομπή μικρότερη από 70 γραμμάρια. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Βιντάλ Κουάδρας που είπε για τη δημιουργία κινήτρων για να αγοράζουν τον αυτοκίνητο. Αυτό δεν μπόρεσα να το συμπεριλάβω εγώ, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, τι γίνεται σε κάθε επίπεδο ε, και τοπικής αυτοδίκης και σε όλα τα επίπεδα ως βέλτιστη πρακτική. Και ξέρουμε ότι σιγά σιγά χρησιμοποιούνται και λιγότερο ρηπογόνο αυτοκίνητα και τα ηλεκτρικά οχήματα. Σωστό είναι αυτό. Τόσο αναφορά τον ε, κύκλο δοκιμών και την όνισε. Έχω το εξής πρόβλημα. Εμείς ε, που παίρνουμε τις πολιτικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα πρέπει να νύπτω με τα χείρα μας και να λέμε ότι όλα αυτά τα αφήνουμε σε αυτή την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών να αποφασίσει. Εμεί είμαστε υπεύθυνοι γιατί γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, όπω είπε και η Επιτροπή, τον κύκλο δοκιμών. Είμαστε λοιπόν υπεύθυνοι και θα πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση και προσαρμογή και όπω είπε και η Επιτροπή συνακτικά είμαστε σε θέση να κάνουμε ε, τις διάφορες αναπροσαρμογές όταν θα εμφανιστεί και η έκθεση Ιονισή. Δεν θα πρέπει όμως να νύπτουμε τα χείρες μας, διότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Είμαστε υπεύθυνοι ως πολιτικοί και πρέπει να υπομισθούμε την ευθύνη μας. Και τελικά κάτι για τον κύριο Κράμερ. Εδώ Μιλούμε για τον κανονισμό που αφορά τις εκπομπές εξουσίου του άνθρωπος για τα ε, αυτοκίνητα. Πρόκειται όχι για το σφαιρικό πρόβλημα, ένα μέρος του προβλήματος. Βεβαίως υπάρχουν κι άλλα εκτός αυτού. Δεν θα πρέπει όμως να τη συγχαίουμε θα πρέπει αυτό το κανονισμό που εξετάζουμε τώρα να είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε ώστε να δουλεύει αποδοτικά. Ευχαριστώ την κυρία Χολ. Η προθεσμία κατά τροπολογιών είναι 31 Ιανουαρίου το μεσημέρι και η ψηφοφορία προβλέπεται για την 19 Μαρτίου τώρα σε ό,τι αφορά την πρόταση που είχε κάνει ο Βιδαλ Κουάντρος για τον ε, συνδυασμό των συζητήσεων επί των δύο εκθέσεων. Το μοναδικό πράγμα που έχουμε ανάγκη είναι ότι θα ήταν ενδιαφέρον και χρήσιμο να πετύχουμε συμφωνία οι δύο εισηγητέ, η κυρία Χόρ και ο κύριος Πίπερ. Σας υπενθυμίζω ότι στις 11 θα έρθει ο Ιρλανδός Υπουργός, ο κύριος Ράμπιτ, Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαι πολύ αυστηρή με τον χρόνο. Ζητώ συγγνώμη, καθυστερήσαμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα. Αφορά στην προστασία των φυσικών προσωπών ε, έναντι επεξεργασία δεδομένων, προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων, ο συνάδελφο Κέλλη έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα μου χρειαστούν πέντε λεπτά. διότι ο χρόνος πιέζει. Να πω πως ο κανονισμός περνάει σε μια κρίσιμη φάση συζητήσεων. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Έγινε συζητήσει ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες και θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε αντανακλά τα ζητήματα που έθιξε και ο κ. Πίπερ και η κυρία Χολ ε, σχετικά με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του κανονισμού όπως αυτός προτείνεται από την Κομισιόν και δυστυχώς κάποιες από τις προτάσεις που έρχονται από τον ε, κύριο Άρμπεχτ και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ε, ε, η εκτίμηση μάλλον αντικτύπου που υποβλήθηκε πριν από τα Χριστούγεννα αγνοήθηκε και αυτό όμως θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη διότι είναι απογοητευτικό να παρατηρούμε ότι πολλοί θεωρούν πως αν επιθυμείτε να προστατεύσετε τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορείτε να ε, προστατεύετε και τους ε, καταναλωτές. Αλλά στην ουσία πρόκειται για το αυτό ζήτημα. Εμείς αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται να εξετάσουμε πώ η νομοθεσία μπορεί να επηρεάζει την βιομηχανίε ειδικά στην Ευρώπη. Ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας έχουμε νομίζω την υποχρέωση σε αυτή, ειδικά την Επιτροπή, να εξετάσουμε τις ανάγκες και τις ανησυχίες των βιομηχανιών. Όλα αυτά τα έλαβα υπόψη μου στις τροπολογίες. Ε, θα ήθελα απλά να αναφέρω κάποιες από αυτές. Αν έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, παρακαλώ να με, κόψετε, να με διακόψετε. Στη τροπολογία στο άρθρο 2 είναι πολύ σημαντικό διότι αποτελεί μια διευκρίνηση του πεδίου εφαρμογή. Επίση, ο ορισμό του ελεκτή και αυτή η αποσαφήνιση νομίζω ότι είναι χρήσιμη. Χθε είχα μια συζήτηση, τρεις συναντήσεις με οι ηγητές οργανώθηκαν, έλαβαν χώρα χθε. Προσπαθούμε να πετύχουμε συμφωνία σχετικά με 77 συμβαστικές τοπολογίες, αλλά ακόμα πολλές συζητήσεις πρέπει να διεξαχθούν στο ενδιάμεσο. Επίσης ε, υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω. Έχω τροπολογήσει. A focus on Και η απλούστευση της ε, Όλη η διαδικασία ε, που αφορά στο άρθρο 26 διαγράφηκε διότι δεν προσέφερε κάποια διευκρίνηση. Επίσης ε, έχω την τροπολογία υπερθμών 26 που μιλάει για την ε, ψευδονιμοποίηση. Το νέο άρθρο 33 που την, προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. Άρθρο 33, παράγραφος 1 ε, για τις εξαιρέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ε, της λειτουργίας ε, της προστασίας δεδομένων και για την περίοδο αυτής νομίζω ότι με την εξάρτηση από τη συγκατάθεση. Επιθυμούμε επίσης να μειώσουμε την γραφειοκρατία για την προηγούμενη διαβούλευση, η οποία δεν θεωρώ ότι απαιτείται σε κάποιους τομείς. Άρθρο 39 και για την διεθνή μεταφορά δεδομένων, να αναφέρω το άρθρο 42, για τους ε, διαχειριστές ε, αυτών των δεδομένων το θέμα της συμμόρφωσης Ο χρόνος ε, έχει περάσει όμως, άλλες δύο, ε, άλλα δύο άρθρα, άρθρο 58, ζητάω να διαγραφεί. Και το άρθρο 60 και εδώ διαγραφή. Έλ, έληξε ο χρόνος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Τικάου έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Κέλλη για την συνεργασία που είχαμε ήδη η Μεστερία ιδιαίτερα φορτωμένη με τις συναντήσεις των σκιωδών ε, χθες είχαμε μια ώρη συνάντηση, ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και αποδοτική. Σε ό,τι φορά τις τροπολογίες θα στηρίξουμε όλες τις τροπολογίες που περιορίζουν το δικαίωμα της Επιτροπής να παρεμβαίνει μέσω των πράξεων κατά την εξουσιοδότηση. Ε, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της τεχνολογικής ουδετερότητας, privacy by design και privacy by default, ε, εξσχεδιασμού. Επίσης ε, δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αυστηροί, θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις και ειδικά στις, μικρο, στις μικρές, ενώ δεν ε, ισχύουν για τα ευρωπαϊκά όργανα που επεξεργάζονται στοιχεία προσωπικά δεδομένα. Επίσης ε, υπάρχουν και ε, ε, κάποιες τροπολογίες που φορούν την περαιτέρω διευκρίνηση κάποιων ορισμών. Χθε μιλήσαμε για τα ανανυμοποίηση και για τα την ψευδονυμοποίηση, αλλά όπως είπε και ο εισηγητής, θα είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια επόμενη συζήτηση πολύ πιο ε, ενδελεχής, διότι εδώ μιλάμε για ουσιώδη δυσδήματα. Και κάτι ακόμα που αφορά τις διεθνείς συνθήκες. Εμείς μέσω των τροπολογιών μας θελήσαμε να ορίσουμε μια μεταβατική περίοδο πενταετή. Προτού η οι διεθνείς συνθήκες τεθούν σε εφαρμογή, αλλά ήδη ξεκίνησαν διαπραγματεύσει για την προσαρμογή αυτών των διεθνών συμφωνιών. Και θα επηρεάσουν και τα ευρωπαϊκά δεδομένα και το σχετικονισμούς. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί ιδιαίτερα σημαντικοί, όπως το ζήτημα της, ε, των μητρών επιβατών αυτό θυμάστε ότι είχε προκαλέσει μια σειρά συζητήσεων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νομοθεσία που θα εφαρμοστεί στον τομέα. Αναφέρουμε στα δεδομένα τα οποία τυχαίνουν χάνουν σε διεθνές επίπεδο. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν θα πρέπει να έχουμε έναν κανονισμό ε, ε πιο αδύναμο από τη μία οδηγία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ενεργήσαμε καταλήλως. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτή η συνένεση, αυτή η συγκατάθεση θα δίνεται με τρόπο ενημερωμένο, με έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Τώρα σημαντικά είναι για τα στοιχεία των πολιτών τώρα. Σε ό,τι αφορά την χρονική περίοδο, ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν, αλλά προτείνουμε 72 ώρες αντί 28 για την διαγραφή. Είμαι πεπισμένη ότι θα συνεργαστούμε άψογα με τον συγητή. Ε, ο κανονισμός είναι απλός, μη γραφειοκρατικός, εύκολος στην εφαρμογή του και ιδιαίτερα σημαντικός για τους πολίτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> Και εμείς από την ομάδα μου καταθέσαμε με τους συναδέλφους κάποιες τροπολογίες ώστε να υπάρχει ευελιξία και προστασία των δεδομένων σε αυτό τον κανονισμό. Θέλησαμε να υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και την συνένεση σαφής ορισμός λέγοντας ότι ότι τα δεδομένα που αφορούν ατομικά κάποιον αφορούν αυτόν τον κανονισμό και οι συνένεση θα πρέπει να είναι σαφής χωρίς αμφισημίες. Τώρα, θέλουμε ο ελεγκτής να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει έναν εκπρόσωπο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επεφεληθεί από το One Stop Shop. Επίσης, θελήσαμε την προστασία των δεδομένων να την διαχωρίσουμε από άλλα θέματα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με την νομοθεσία των κρατών μελών. Πιστεύουμε ούτως ή άλλως ότι κάποιοι ειδικοί τομεί μεταξύ των οποίων κάποιοι είναι τομείς στους οποίου υπάρχουν πάρα πολλοί κανονισμοί, δεν θα πρέπει να υποστούν από αυτόν τον κανονισμό πολύ περισσότερο άχθος. Επίσης, καθορίσαμε το ρόλο και τις ευθύνες των, ε, αυτών που επεξεργάζονται και ελέγχουν τα δεδομένα και είπαμε ότι οι ελεγκτές των δεδομένων θα πρέπει να ασχολούνται θεωρητικά με το θέμα αυτό και επεξεργαστείς με τα διαδικασίες της ε, εκτίμηση θα πρέπει να την κάνουν οι ελεγκτές. Είπαμε ότι θα πρέπει να ξέρουν οι ΜΜΕ. Πρώτα απ' όλα για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πρέπει να ορίσουν έναν πρόσωπό τους για την ε, προσία των δεδομένων ή να κάνουν μία ε, μελέτη προστασίας της ιδιωτικής ζωής τις τρία πρώτα χρόνια των δραστηριοτήτων. Ε, θα πρέπει αναμφίβολα θα πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ώστε να προστατεύουμε τα δεδομένα της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό και θα πρέπει να κάνουμε νομοθεσία η οποία δεν θα βοηθήσει την ε, προστασία των προσωπικών ε, δεδομένων, αλλά θα δημιουργήσει περαιτέρω οικονομικά προβλήματα και δυναμίες στις ε, εταιρείε μας και στις διάφορες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντερς Ντότερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή μας ξέρουμε ότι έχει ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ε, βιομηχανίες και έρευνας. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει σήμερα να κάνουμε κάτι διαφορετικό όλο και περισσότερο. Θα πρέπει εμείς να έχουμε ηγετικό ρόλο για την βιομηχανία και να βοηθήσουμε και τις ΜΜΕ θα πρέπει να διατηρηθεί το επίπεδο προστασίας των δεδομένων των πολιτών μας όπως κάναμε τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε κάνει εκτενείς έρευνες για να ξέρουμε πώς εφαρμόζεται το θέμα. Έχουμε έρευνα από τα πανεπιστήμια και ξέρουμε ότι και σε επίπεδο εθνικό έχουμε εμπειρία. Χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη προστασία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να υπάρχει πάντα σωστή εφαρμογή σε όλα τα κράτη δικαίου. Ξέρω ότι πολλές χώρες ξέρουν τι γίνεται όταν ε, κάποιος ε, καταχράται αυτό το σύστημα προστασία των δεδομένων. Θέλουμε στις κοινωνίες μας να είναι δημοκρατικές. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην προσωπική του ζωή, στην δική του ζωή και στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Όταν μιλάω εγώ σε για το πώς μπορούμε στον τομέα αυτό να βελτιώσουμε την ε, πολιτική μας, πολλοί μου λένε ότι εμείς έχουμε σηκώσει τα χέρια, δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο και κανένας δεν μπορεί να τους το προσάπει αυτό. Σήμερα όμως έχουμε εκθέσεις, έχουμε επιστημονικά δεδομένα, έχουμε τις ε, σχετικές ε, ρυθμιστικές αρχές σε κάθε χώρα, το άρθρο 29, γι' αυτό ζητούμε την Επιτροπή να μελετήσει το θέμα αυτό καλύτερα, ώστε το πλαίσιο προστασίας δεδομένων να μπορέσει εθνικό, διεθνές ε, ε, επίπεδο είναι ανταγωνιστική. Έχουμε πολλές εκατοντάδες τροπολογιών που πολλές ε, είναι αρνητικές και αν εγκριθούν θα γίνουν ε, θα υπάρξει τρομερό πρόβλημα και για την βιομηχανία και για τους ιδιώτες. Θα δημιουργηθεί λοιπόν μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε το επίπεδο προστασίας που είχαμε το 1995 είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε και αυτός είναι ο ελάχιστος στόχος που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όλους τους συναδέλφους ώστε να διαδραματίσετε τον ρόλο που διαδραματίσατε ως τώρα και ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αποτύχουμε. Δεν ήρθε η κατάλληλη στιγμή να υποχωρήσουμε, αλλά να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προς τη στόντη κατεύθυνση, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο επιθυμούν οι πολίτες μας και έχουν το δικαίωμα να το απαιτήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο, ο κύριος Τσίτσεστερ έχει το λόγο. Um, thank you, Madam Chairman. Uh, I thought I was going to help your εγώ είχα σκεφτεί μήπως να μην μιλήσω για να προλάβουμε καλύτερα. Υποστηρίζω, γι' αυτό θα πω μονάχα, τον εισηγητή και την καλή δουλειά που έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε χρόνο πολύ. Δεν θα είμαι το σύντομο ο συνάδελφος Τσίσεστερ, αλλά σύντομη αρκετά στην παρέμβασή μου. Πιστεύω ότι ο λόγος ύπαρξης αυτής της πρότασης αναθεώρησης για την προστασία των δεδομένων έχει στενή σχέση με τις ε, μεταβολές που έχουμε εξαιτία της ψηφιακής κοινωνίας στην οποία ζούμε. Και πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος αυτά που είπε και τον προσανατολισμό που παίρνει, διότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Φερρυπίν, όπως ανέφερε, και αυτό είναι ένα σύνηθες θέμα όταν συζητήσουμε τις ε, αρμοδιότητες, την ευθύνη του επεξεργαστή και του ελέγχτη των δεδομένων. Άρα με αυτή την έννοια η πρόταση της Επιτροπής πιστεύω ότι παρά την ε, καλή της βούληση δημιουργεί κάποια σύγχυση όσον αφορά τις ευθύνες. Νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής μας μέσω του κυρίου Κέλλη και με τις ε, προτάσεις των σκιωδών ε, εισηγητών θα μας βοηθήσει από την Ήτρε να υπάρχει μία συνεισφορά που θα βοηθήσει στο να αποσαφινιστούν κάποια θέματα. Δηλαδή, ποιοι είναι τόσο σημαντικοί στην ψηφιακή μας ε, κοινωνία σήμερα, χωρίς να υποστεί πλήγμα ο δυναμισμός των νέων τεχνολογιών της ψηφιακής κοινωνίας και του ίντερνετ. Είναι θεμελιώδη σημασία η καινοτομία, πρόκειται για πολύ δυναμική τεχνολογία της οποίες δεν θα μπορέσουμε να καταστήλουμε από κανονισμούς που θα δημιουργήσουν ασφυξία και στην πράξη ούτως ή άλλως δεν θα είναι χρήσιμες, δεδομένου ότι η τεχνολογία προχωρά πολύ πιο γρήγορα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ ισοσκελισμένη πρόταση. Τη συζητήσαμε δύο, τρεις, τέσσερις και παραπάνω φορές στην Επιτροπή μας. Απλώς και μόνο θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία που επιτέλεσε, που κατά άποψή μου είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιδάλ Κουάδρας. Κυρία Πρόεδρε, στα πλαίσια της οδηγίας του 95 πρέπει να πω ότι είναι σημαντική, Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την όθηση της τεχνολογίας και τα μεγάλα βήματα που έγιναν από τότε. Η πρόταση της Επιτροπής φτάνει την κατάλληλη στιγμή και ελπίζω ότι θα οδηγήσει σε εναρμόνιση της προσίας των δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εφησυχάσει όλους αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Κέλλη για την εργασία που επιτέλεσε για την γνωμοδότηση αυτή και κυρίως συμφωνώ με το στόχο του να μειωθεί το διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις και να μην επιτρέψει στην οικονομική ανάπτυξη να ε, έχει προβλήματα εξαιτήματα της υπερβολικής γραφειοκρατίας όσον αφορά τον ελεκτή και τον επεξεργαστή δεδομένο, Προτείνει να αναπαιτείται ότι κάνουν, να το κάνουν στα πλαίσια αυτού του κανονισμού. Και όχι ότι κάνουν να το κάνουν με στόχο να αυξηθεί ο φόρτος εργασίας που έχουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα με λογική, φέρει οι επιχειρήσεις μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να προστατεύονται από τις απάτες, για να φέρω ένα παράδειγμα, για να μπορέσουν ε, να κάνουν ε, συστάσεις αποδοτικές και για άλλους. Ε, η ψευδονιμοποίηση και η ανωνυμοποίηση των δεδομένων μπορούν να είναι κάτι το πολύ χρήσιμο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα πρέπει να γίνονται εκθέσεις αναφοράς και να μην γίνονται καταχρήσεις. Καλή δουλειά κάνατε κύριε Κέλλη. Θα σας υποστηρίξουμε. Επιτροπή παρακαλώ. Έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομος. η Κομισιόν αναμένει με ενδιαφέρον τις τροπολογίες. Χρειαζόμαστε ρύθμιση ασφαλή για το μέλλον για τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους, εις τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί ο υψηλότερος βαθμός προστασίας για τα πρόσωπα, αλλά ταυτόχρονα να διατηρηθεί και περιθώριο κίνησης για τις επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν. Η Κομισιόν σε κάθε προσπάθεια αποφυγής της γραφειοκρατίας συμπαρατάσσεται και αυτό είναι, αυτή είναι η έννοια των ρυθμισιών μας. Από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. ώστε οι ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων να είναι καλές και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να μην προκαλούν να μην έρχονται αντίθετες οι διατάξεις προστασίας των δεδομένων για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντίθετα να είναι προϋπόθεση. Χωρίς προσωπικά δεδομένα και ιδίω για την ψηφιακή ατζέντα δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Οι πολίτες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι η οικονομία, η βιομηχανία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα με τον πρέποντα τρόπο. Η Κομισιόν προσπάθησε προσπαθεί να διατηρήσει και να βελτιώσει την προστασία που προσφέρει η Οδηγία 9546 και να μην μειωθεί το επίπεδο αυτό προστασίας. Θα εξετάσουμε λοιπόν με μεγάλη προσοχή τις τροπολογίες που θα υποβληθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Για πέντε λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όλες και όλους. Όσα άκουσα ήταν και ειλικρινή και σημαντικά. Άκουσα κάτι περί σύγχυσης στην αρχή. Έχουμε χρέος να ξεδιαλύνουμε οποιαδήποτε σύγχυση. Όπου θίγονται οι καταναλωτές, δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση σχετικά με τα δεδομένα τα οποία κάπου αποθηκεύονται για το άτομό τους. Η λύση δεν είναι απαραίτητα περισσότερη ε, νομοθεσία, αλλά καλύτερη ποιοτικά. να είναι εξασφαλισμένα τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών και ιδίω. αυτή η όλο και αυξανόμενη σιωπηρή συνένεση πρέπει να αντιμετωπιστεί γιατί υπάρχει και αυτή η κόποση του κλικ όπως λέγεται. Δηλαδή κάποια στιγμή ο καταναλωτής δεν θέλει πλέον να πατάει κουμπιά για να λέει ότι δεν θέλει να διοχετεύονται παραπέρα τα δεδομένα του. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε το επίπεδο προστασίας, όπως είπε και η Κομισιόν, για, με τη σχετική οδηγία, αλλά να καταστεί επίσης σαφές, αλλά και να είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ε, το σχετικό σύνολο ρυθμίσεων. Νομίζω η Σίλβια είπε για τις κατεξουσιώτηση πράξεις. Εμείς θέλουμε να τις μειώσουμε αυτές, στο ελάχιστο δυνατό. Γιατί πολλές κατεξουσιώδει πράξει σημαίνει ότι καταρχήν, ο καταρχήν σχεδιασμό τη ρύθμιση δεν ήταν επαρκή. Επίση, η μοναδική, η ενιαία θηρίδα, το One Stop Shop, είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πολλές επιχειρήσεις. Είναι κρίσιμο εάν θέλει κανείς να έχει πανευρωπαϊκή ρύθμιση. Αυτό το One Stop Shop είναι απόλυτα λογικό και να μην το αποδυναμώσουμε ώστε να στερείται νοήματος εν τέλει. Και αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Για τον ελεγκτή και χειριστή, εδώ χρειάζεται επίσης αφήνεια για το ποιο είναι ο ελεγκτής που αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη πτυχή, ενώ ο processor άλλη. Αυτό πρέπει να είναι και το modus operandi που θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Μία από τις προτάσεις που προκαλεί πολλές δυσχέρειες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και η ανάγκη ενός εντεταλμένου την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενός DPO, Data Protection Officer. Πολλές επιχειρήσεις ανησυχούν για τη ρύθμιση αυτή. Άρα και εδώ πρέπει να σκεφτούμε κυρίως την πρακτική εφαρμογή και να δούμε και τον όγκο των δεδομένων που ε, χειρίζεται μια ε, επιχείρηση. Λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχει ανάγκη. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων, ανάλογα με το μέγεθός τους. Και αυτό πρέπει να το δούμε λοιπόν. Σήμερα το πρωί ήδη, σε μια ραδιοφωνική ακρόαση για μερικά από για μερικά θέματα όπου ανησυχούν κάποιοι στον τομέα της υγείας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί ο τομέας της υγείας χρησιμοποιεί πολλά, όγκο μεγάλων δεδομένων. Μπορεί να φτάσουμε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου έχουμε ανεπιθύμητες επιπτώσεις και που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον τομέα της υγείας, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε, αυτήν, σε αυτόν. Και αυτά λοιπόν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εν συμπεράσματι, όλοι βέβαια θέλουμε να διατηρήσουμε υψηλή προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων, ταυτόχρονα όμως δεν θέλουμε να παρεμποδίσουμε την ανάπτυξη των μικρών και μεσών επιχειρήσεων που υπάρχουν ήδη, δραστηριοποιούνται και ιδίω βέβαια την καινοτομία που όλοι λέμε πόσο σημαντική είναι για την Ευρώπη. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία. Και αναμένω με ενδιαφέρον τις προτάσεις και απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ολοκλώσαμε αυτό το κομμάτι των εργασιών. Πενθυμίζω ότι 21 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία κατά τροπολογία. έχουμε την... Τώρα θα ακολουθήσει η παρουσία του κυρίου Υπουργού. Όσοι δεν επιθυμούν να παραστούν, παρακαλούνται να αποχωρήσουν τώρα ησύχως. Υπότιτλοι Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας ε, τον Υπουργό Ράμπιτ, Ιρλανδό Υπουργό για τις επικοινωνίες, την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους σου. Εκπροσωπεί την Προεδρία τον ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία του και ευθύ αμέσω του δίνουμε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Madam Chairperson, ε, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, πρώτη τιμή για μένα που μου επιτρέπετε να αναπτύξω το πρόγραμμα της Ιρλανδικής Προεδρίας στην Επιτροπή Βιομηχανίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω ζητήσει πάντοτε εγώ ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έτσι ως υπουργό αλλά και εκλεγμένος βουλευτής του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου γνωρίζω και είμαι πλήρως ενήμερος και εκτιμώ τον κέριο ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην δημοκρατική διαδικασία. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη μιας πιο δημοκρατικής και διαφανούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, εποφελία των πολιτών, είναι ιδιαίτερα σημαντική φέτος που είναι και έτος του πολίτη και μέσα στα πλαίσια βέβαια των θεμάτων της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Η Ιρλανδική Προεδρία αναμένει θετική και επικοδομητική σχέση με το Κοινοβούλιο. Ανά πάσα στιγμή θα κάνουμε προσπάθεια να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς ως Προεδρία. Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα και βέβαια με στόχο τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εκτιμώ ιδιαίτερα την, ε, την γνώση και εμπειρία της Επιτροπής σας και ελπίζω να βασιστούμε σε μια σχέση συνεργασίας την οποία επιζητούμε. Η σχέση αυτή έχει ήδη σφυριλατηθεί από τις προηγούμενες επαφές και συναντήσεις μας μεταξύ, αυτών, μεταξύ άλλων με την κυρία Σαρτόρη καθώς επίσης και την πολύ παραγωγική επίσκεψή σας στο Δουβλίνο. Τα κυρίαρχα θέματα της ε, Προεδρίας μας θα είναι οι τρεις προτεραιότητες σταθερότητα, απασχόληση και ανάπτυξη. Η Ιρλανδία θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι της Ένωσης θα στοχεύουν στα απαραίτητα βήματα για την αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας, απασχόλησης και ανάπτυξης. Ιδιαίτερα θα δώσουμε προτεραιότητα σε ε, πρωτοβουλίες νομικές και πολιτικής για την ενιαία αγορά και για την ψηφιακή ατζέντα. Η ενιαία αγορά έχει αποδώσει πολλά ωφέλη στις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και καταναλωτές. Η Προεδρία μας θέλει να επιτύχει πρόοδο σε εκρεμή θέματα ακόμα από την πρώτη πράξη ενιαίας αγοράς μεταξύ αυτών και την ψηφιακή ενιαία αγορά όπως ήδη περιλαμβάνεται και στο ίδιο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης αναμένουμε τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων με τα μέτρα της νέας πράξεω 2 της ενιαία αγοράς. Εδώ χρειάζεται σημαντική προσπάθεια, ιδίως στη βάση της διευκόλυνση επενδύοντας, ε, συνδέοντας μάλλον την Ευρώπη. Οι τομείς αυτοί δηλαδή μεταφορές ενέργεια και τηλεπικοινωνίες, είναι και στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Η Κυπριακή Προεδρία επέτυχε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κατευθυντήρες γραμμές της ενέργειας. Και εδώ χαιρετίζω τον κύριο Κορέα Ντεκάμπος, εισηγητή. Επίσης, για τις κατευθείαν γραμμές των τηλεπικοινωνιών, που θα είναι μία από τις ε, κέρυες προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Αν και εδώ αυτό, η επιτυχία αυτού του μέτρου θα εξαρτηθεί από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, εμείς ως Προεδρία θεωρούμε ότι η λογική και η δομή του μέτρου δεν πρέπει να εξαρτάται από το ακριβές ποσό των χρημάτων που θα διατεθούν σε αυτό. Η Κυπριακή Προεδρία επέτυχε σημαντική πρόοδο στον ε, φάκελο αυτό. Ωστόσο χρειάζεται περισσότερη δουλειά σε έναν αριθμό τομέων. Η Ιρλανδική Προεδρία θα προσπαθήσει να δώσει τελική μορφή στις απόψεις του Κοινοβουλίου τις οποίες μετά μπορούν να υποστηρίξουν οι χώρες μέλη για να ανοίξουν το δρόμο για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διάβασα με ενδιαφέρον το σχέδιο εκθέσεως του κ. Τοσενόφσκι και σημείωσα ότι τα θέματα που θέτει το Κοινοβούλιο είναι παρόμοια με αυτά που συζητεί το Συμβούλιο. Η, Ευρωπαϊκή, Προεδρία θα προσπαθήσει να δώσει τελική μορφή στις ε, απόψεις του ε, Συμβουλίου και να ανοίξει τον δρόμο για τις ε, συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συναντήσει τον κύριο Τωσενόφσκι σήμερα αργότερα για να αναζητήσω μαζί του τους καλύτερους τρόπους για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό σε πρώτη ανάγνωση. Υπάρχουν άλλοι δύο φάκελοι των τηλεπικοινωνιών μετά από τον τριμερή διάλογο που έχει αρχίσει η Υποκυπριακή Προεδρία. Ο πρώτος είναι πρόταση για την εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Εδώ μπορούν να προκληθούν, ε, να δημιουργηθεί νέα απασχόληση, εφόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιες πληροφορίες με περιθωριακό ή καθόλου κόστος. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα να αναπτυχθούν νέα καινοτόμα από καταναλωτέ αλλά και για τι επιχειρήσει. Και έτσι θα είναι σημαντική η συμβολή προ την κατεύθυνση τη ολοκλήρωση τη ε, ενιαία ψηφιακή αγορά. Μετά από τον πρώτο πολύ επικοδομητικό τριμήρη διάλογο υπό την Κυπριακή Προεδρία. Εγώ σημειώσα ότι το Κοινοβούλιο με την καθοδήγηση του εισηγητού κ. Κάλφιν συμφώνησε με το Συμβούλιο ότι είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Η Ιρλανδική Προεδρία δεσμεύεται να προσπαθήσει να το επιτύχει. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται στην ένισα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών και την πρόταση ενίσχυσης και εξυγχρονισμού του οργανισμού αυτού με νέα εκτεταμένη εντολή για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Γνωρίζουμε όλοι ότι η τρέχουσα εντολή της ένισα εκπνέει σε λίγους μήνες. Η Ιρλανδία ως Προεδρία πιστεύει ότι αναπόκειται και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να επιτύχουν συμφωνία στο φάκελο αυτό, δίνοντας έτσι την απαραίτητη σαφήνεια για το μέλλον της, του οργανισμού ένισα. και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν ότι η ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και η αύξηση στους αριθμούς συμβάντων στον κυβερνοχώρο αλλά και απειλών ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίσιμη αυτή ευρωπαϊκή υποδομή και είναι θέματα τα οποία χρειάζεται άμεση μελέτη. Χαίρομαι λοιπόν για το γεγονό ότι τριμερής διάλογος έχει οργανωθεί για τις επόμενες ημέρες και θα συζητήσω το θέμα αυτό αργότερα σήμερα με τον κύριο Τσίτσεστερ. Άλλωστε έχουμε συναντηθεί με τον κύριο προμηνών. Οι ασφαλείς, αξιόπιστες και εύκολες επιγραμμικές συναλλαγές είναι σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Ο προτινόμενος κανονισμός για ηλεκτρονική ταυτοποίηση και ε, υπηρεσίε εμπιστοσύνη έχει κέρια σημασία. Η Ιρλανδία γνωρίζει τη σημασία αυτού του κανονισμού αλλά καθώς επίσης και την περιπλοκότητά του συμμετέσχουν πρόσφατα σε Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών και άκουσα εκεί και τις ανησυχίες των Υπουργών. Για μένα κατέστη σαφές ότι απαιτείται πολύ και λεπτομερή εργασία για ορισμένα θέματα, αλλά με ενθάρρυνε η ευρεία υποστήριξη που δίνεται στην πρόταση. Εγώ βεβαίωσα τους Υπουργούς ότι η Προεδρία θα εργαστεί για να κάνει την ε, οδηγία αποτελεσματική όσο γίνεται περισσότερο. Για τον για το Συμβούλιο του Ιουνίου θα έχουμε μια progress report για να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις αργότερα. Χαίρομαι για την ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή σας και γνωρίζω ότι έχουν τεθεί και τέτοια θέματα. Στην ψηφοφορία σας του Ιουλίου η φιλοδοξία μου είναι η θέση του Συμβουλίου να έχει προχωρήσει. Η σημασία των, της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών είναι και προϋπόθεση για να ανθίσει η ψηφιακή αγορά. Και αυτό είναι ένα θέμα για την επικείμενη στρατηγική για την ε, κυβερνοασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει σύντομα τη στρατηγική αυτή μαζί και με σχετική νομοθετική πρόταση. Η Προεδρία θα εργαστεί για να επιτύχει σημαντική πρόοδο για την νομοθεσία αυτή. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας επιχειρήσεων και καταναλωτών αντίστοιχα για να αυξηθεί η επιγραμμική ανάπτυξη. Οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να παράσσονται μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής υποδομή. Η ταχεία ανάπτυξη δικτύων ευρέως φάσματος μεγάλης ταχύτητας είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση. Εμείς κατανοούμε εμείς ε, ε, γνωρίζουμε μάλλον ότι η Κομισιόν θα υποβάλει σχετική πρόταση στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Η Ιρλανδία δημοσίευσε την στρατηγική της, την εθνική της στρατηγική για το ευρύ φάσμα τον Αύγουστο του 2012 και αυτό μας επέτρεψε να αντιληφθούμε ποιες είναι οι προκλήσεις της μείωσης των φραγμών για την ανάπτυξη του ευρώ φάσματος. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την πρόταση της Κομισιόν και θα ηγηθούμε μιας σε βάθος συζήτησης. Θα αρχίσουμε επίσης να εξετάζουμε την πρόσφατα δημοσιευθήσα πρόσφαση, ε, πρόταση μάλλον για την προσβασιμότητα στο δίκτυο σημαντική πρόταση αυτή, ιδίω για το 2013, που είναι ε, το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών. Το έργο της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι και επίκαιρο, διότι πρόσφατα δημοσίευσε η Κομισιόν την mid-term review για την στρατηγική της ε, ψηφιακής ατζέντα. Πρέπει αυτή η φιλοδοξία να διατηρηθεί, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταγωνιστούμε διεθνώς την ε, Επίτροπο κυρία Κρούς ότι η προσπάθεια μας αυτή θα είναι διαρκής. Αυτή η επανεξέταση θα αποτελέσει και την βάση για τις εργασίες της συνέλευσης ε, ψηφιακής ατζέντα που θα γίνει το, στο Δουβλίνο τον επόμενο Ιούνιο και ελπίζω να δω εκεί και πολλού ευρωβουλευτέ. Η Ιρλανδική Προεδρία συνεργάζεται με την Κομισιόν για την διοργάνωση τη εκδήλωση αυτή. Ω Υπουργό Αρμόδιο και για την ενέργεια και για τις ε, τηλεπικοινωνίες με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συνέργειες μεταξύ των δύο τομέων. Αναμένουμε τον Απρίλιο την δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις τεχνολογίες ενέργειας και στα πλαίσια της μελλοντική ευρωπαϊκής πολιτικής της ενέργειας. Σε, ε, στο πλαίσιο βέβαια των προτεραιοτήτων του 2020, την μείωση χρήσεως ε, των καυσίμων για ε, τον οδικό χάρτη 2050 και το σχέδιο ΣΕΤ. Οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν την ανακοίνωση αυτή στο Λουξεμβούργο τον Ιούνιο στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Η πρόοδος της εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι σημαντική για την ανάπτυξη των στόχων ενέργειας της Ευρώπης. Και βεβαίως για να ωφεληθούν και οι καταναλωτές και τα ε, ε, νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Χρειάζεται λοιπόν η μέγιστη πολιτική ορατότητα και βεβαίω αυτό θα το κάνουμε τον Φεβρουάριο στο Συμβούλιο της Ενέργειας, οι εργασίες του οποίου θα τροφοδοτήσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαΐου για το θέμα της ενέργειας. Θα υποβάλουμε συγκεκριμένα πορίσματα του Συμβουλίου συμπεράσματα βάλουν του Συμβουλίου στον Ιούνιο για να τα εγκρίνουν οι Υπουργοί. Η εσωτερική αγορά ενέργειας μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό και αναμένω τις απόψεις της Επιτροπής σας για την ανακοίνωση και βεβαίως ιδίως τα σχέδια του καθηγητού Μπούσεκ για την συγγραφή εκθέσεως για την πρόταση αυτή. Μετά από τη σημαντική πρόοδο που επετέλεσε η Κυπριακή Προεδρία, ο στόχος μας για την πρόταση για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εξόριξης πετρελαίου και φυσικού αερίου θα τεθεί υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιθανώς πριν από το Συμβούλιο Ενέργειας της 22ης Δευτέρου. Ήδη έχω συζητήσει ε, τον προηγούμενο Μάιο με τον εισηγητή σας κύριο Ιβο Μπέλετ και συμφωνήσαμε ότι μπορούμε να τα βρούμε. Ένας κέριος στόχος για την ενέργεια της Ευρώπης είναι η μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, η ανάπτυξη καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, ασφάλεια ενέργεια και ποιότητα περιβάλλοντο. Οι ανανεώσιμε ενέργειε θα παίξουν κέριο ρόλο στην διαμόρφωση του συνδυασμένου, του μέλλοντό μα μάλλον των συνδυασμένων ενεργειών και τη μειώση χρήση του άνθρακα. Η πρόσφατα δημοσιευθήσα οδηγία για την έμεση αλλαγή χρήση γη και την χρήση βιοκαυσίμων και, και βιοϊγρών είναι περίπλοκη πρόταση η οποία περιλαμβάνει και αναφέρεται σε πολλούς τομείς ε, πολιτικής και αφορά κυρίως την μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και χρήση βιοκαυσίμων, καθώς επίσης και τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειές τους στην ε, τοπική παραγωγή ε, τροφίμων. Αυτά αφορούν βεβαίως και τα συμβούλια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, το πρώτο ενέργεια στο δεύτερο περιβάλλοντος και θα υποβάλουμε progress πόρθια για τα δύο συμβούλια τον Ιούνιο που πιστεύουμε ότι θα προσφέρει στην Λιθουανική πλέον Προεδρία που θα μας διαδεχτεί τη στέρεα βάση για τις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζί με τις ανησυχίες για την βιωσιμότητα για τα υγρά βιοκαύσιμα πρέπει να εξετάσουμε και την βιωσιμότητα της βιομάζας γενικότερα. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας, η Κομισιόν αναμένεται να υποβάλει πρόταση οδηγίας για τα κριτήρια βιωσιμότητας της βιομάζας εμείς θα προωθήσουμε τις συζητήσεις αυτές ενεργά. Επίσης θα αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και guidance papers για τις ανανεώσιμες ενέργειες και την στήριξη των σχετικών συστημάτων για τους μηχανισμούς συνεργασίας που προβλέπονται ήδη στην σχετική οδηγία του 2009. Στο δεύτερο μισό της Προεδρίας μας, αυτά θα γίνουν εκεί τότε λοιπόν. Αλλά σημειώνω τώρα με ενδιαφέρον το σχέδιο εκθέσεως του κυρίου Ρόιλ που αναμένει που αναφέρει συγγνώμη, τα δύο αυτά θέματα. Και αναμένω συνεργασία και των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων ενεργειών. Άλλη μείζον προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας θα είναι το δυναμικό των αλλαγών της τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους της του 2020 για την αποδοτική χρήση της ενέργειας. Συγχαίρω τον κύριο Τούρμες για την εργασία που έχει κάνει για την ε, η υποεθανική προεδρία μάλιστα, για την οδηγία αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας. Εδώ χρειάζεται βέβαια αύξηση του ρυθμού της κλίμακας και του βάθους των επενδύσεων, να αναβαθμιστούν τα οι εφιστάμενες εγκαταστάσεις στις χώρες μέλη, για να μπορέσουν έτσι οι χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν σωστά τους στόχους τους για την αύξηση της αποδοτικότητας της ενέργειας. Η χρήση των εφιών συστημάτων, ιδίως εφιών δικτύων και εφιών μετρητών, θα μας στηρίξουν στο μέλλον για την ε, πολιτική μας της ενέργειας και θα συζητήσουμε τα σχετικά στο άτυπο ε, Συμβούλιο Υπουργών τον Απρίλιο, στο Δουβλίνο. Η Προεδρία μας αποδίδει μεγάλη σημασία και στις εξωτερικές σχέσεις ενέργειας της Ένωσης. Στη διαμόρφωση της πολιτικής μας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε σταθερές και διαφανείς παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με άλλους εταίρους για να βάλει τα θεμέλια για μια αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση της ενέργειας. Ωστόσο πρέπει να εμφανιστούμε ενιαίοι, ενωμένοι, ώστε να μεγιστοποιήσουμε το πλεονέκτημα το οποίο διαθέτουμε. Και γι' αυτό χαίρομαι και για την έκθεση του κ. Χέρτσοκ για την εξωτερική συνεργασία ενέργειας. Εμείς θα διερευνήσουμε κέριους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα χρήση της καθαρής ενέργειας για να αυξηθεί η οικονομική ε, δραστηριότητα και η απασχόληση και ούτω Επίσης, αναμένουμε συζήτηση για τι διάφορες πτυχές της διεθνούς συνεργασίας για θέματα ενέργειας στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργεια του Ιουνίου. Στο χαρτοφυλάκιό μου δεν περιλαμβάνονται θέματα πυρηνική ενέργεια, ούτε επίση στο Συμβούλιο. Ωστόσο, το Συμβούλιο ε, Υπουργών Ενέργειας του Ιουνίου θα επιτρέψει στον Επίτροπο κ. Έτινγκερ να ενημερώσει τους Υπουργούς Ενέργειας για τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Οι εκθέσεις του κ. Τσίτσεστερ για τον ε, παροπλισμό ορισμένων, ορισμένων ε, πυρηνικών εγκαταστάσεων και του κ. Κράμερ για την ασφάλεια θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Και θα γίνει και ειδικό συμβούλιο στις 22 Μαΐου για να συζητηθεί ενέργεια δείχνει αυτό πόσο κέρια σημασία θεωρούμε ότι έχει η πολιτική της ενέργειας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτά είναι η υπευθυνότητα του κυρίου Βαν Ρόμποϊ. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα συντήθουν. Ως πρόεδρος της Επιτροπής, ε, ως πρόεδρος, συγγνώμη, του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας θα βάλουμε τον δρόμο για τις συζητήσεις αυτές στο μέλλον. Πριν να ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω τι διοργανώνει η ε, Προεδρία μας φέτος. Το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας τον Απρίλιο. Την σύσκεψη SET Plan τον Μάιο. Επίσης την συνέλευση της ψηφιακής ατζέντα τον Ιούνιο. Και όπως είπα, ελπίζω να δω και μέλη της Επιτροπής σας στις ε, εκδηλώσεις αυτές. Εν συμπεράσματι, το πρόγραμμά μας είναι φιλόδοξο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε σημαντικά και διαρκώς στον κοινό στόχο μιας δημιουργίας, της δημιουργίας μιας ικανότητας που να είναι ψηφιακά ικανή. Και για την πλευρά της ενέργειας θα προχωρήσουμε στο να βάλουμε τα θεμέλια μιας ολοκληρωμένης και διασυνδεμένης εσωτερικής αγοράς της ενέργειας που να εξασφαλίζει την απασχόληση, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα να προστατεύει το περιβάλλον. Και όχι μόνο μέχρι το 2020, αλλά και πέραν αυτό, μέχρι το 2030 και μέχρι το 2050 με τον απότερο στόχο της οικονομίας που θα είναι απαλλαγμένη όσο είναι το δυνατόν αυτό από τα ορυκτά καύσιμα που παράγουν ε, οξύδια του άνθρακα. Και αναμένω βεβαίως τη συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής σας και την στήριξή σας. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Περνάμε τώρα στον πρώτο γύρο των παρεμβάσεων από πλευράς πολιτικών ομάδων. Θα λάβουμε μετά μια απάντηση από τον κύριο Υπουργό και θα συνεχίσουμε. Κυρία Καστίγιο έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλώς όριζατε κύριε Υπουργέ. Είχαμε την ευκαιρία να σας συναντήσουμε στο Δουβλίνο σε μια επίσκεψη που διοργάνωσε η Επιτροπή μας αλλά και σε κάποια άλλη στιγμή εδώ στις Βρυξέλλες πριν ε, από την ανάληψη της Προεδρίας ε, από την Ιρλανδική κυβέρνηση. Καταρχάς να σας πω ότι σε αυτήν την Επιτροπή όπως και πάντα εξάλλου θα δείτε ότι θα είμαστε πάντα διαθέσιμοι, ανοιχτοί, να συνεργαστούμε σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν και για τα οποία εσείς ε, είστε υπεύθυνος ε, κάνατε μια, μάλλον διατρέξατε τα διάφορα ζητήματα με ζητήματα τα οποία θα εξεταστούν κατά την ε, Προεδρία σας, ε, να πω ότι πρόκειται για νομοθετικά ζητήματα ως επιτοπλίστων, διότι πολλά έχουν και την ε, σημασία τους και αφορούν φακέλους οι οποίοι θα συμβάλλουν στο να αναπτύξουμε στρατηγικές μακροπρόθεσμες είναι θέματα πολύ σημαντικά όπως η ιστορική αγορά ενέργειας αλλά και άλλα θέματα. Σε ό,τι αφορά τα νομοθετικά ζητήματα που αφορούν τους στο συγκεκριμένο εξάμεινο της Ιρλανδικής Προεδρίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Φυσικά υπάρχει το Connecting Europe Facility και όλες οι σχετικές υποδομές που θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε νέα δίκτυα, δίκτυα νέας γενιάς και θα βελτιώσουν την ταχύτητα μετάδοσης Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα να σας πω να ασχοληθείτε ιδιαίτερα διότι υπάρχει κίνδυνος να ε, γίνουν πολλές θυσίες ε, στον ε, τομέα των υποδομών για τις τηλεπικοινωνίες. τηλεπικοινωνίες. Δεν θα πρέπει να δοθεί λιγότερη σημασία σε σχέση με την ενέργεια και τις μεταφορές στο ζήτημα αυτό από πλευρά Ιταλική Προεδρία, λοιπόν, θα πρέπει να καταβληθεί μια προσπάθεια η οποία θα εκτιμηθεί διόντω. Ε, ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί το ε, εξάμεινο αυτό. Και, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στι αρμοδιότητέ σα, αλλά είναι αρμοδιότητε τη δική μα Επιτροπή που αφορούν την ψηφιακή κοινότητα αλλά και την ενέργεια και συγκεκριμένα δύο. Πρώτον, η ηλεκτρονική πιστοποίηση που συνδέεται με πολλές από τις πτυχές που εσείς αναφέρατε για την ανάπτυξη της ε, ψηφιακής αγοράς κλπ. Αλλά είναι και ζήτημα το οποίο βρίσκεται επιτάπητος και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η πρόταση της Κομισιόν για τα δικαιώματα εκπομπών. Κάτι το οποίο δεν υπαστεί θα έλεγα ανάμεσα στις Επιτροπές Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος, αλλά αρμόδιοι είμαστε εμείς ως Επιτροπή Βιομηχανίας. Αλλά και σήμερα ο συνάδελφός σας Υπουργός Βιομηχανίας θα μας επισκεφτεί και θα το εξετάσουμε. Πάντως πρόκειται για θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν άμεσα στις αρμοδιότητές σας τόσο σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική επιστοποίηση όσο και το backloading για τις επιπτώσεις που έχει τα θέματα που μας απασχολούν. Θα ήθελα λοιπόν να του αποδώσετε την ε, κατάλληλη τη δέουσα σημασία. Θα έχουμε ευκαιρίες ε, να δούμε πώς θα προχωρήσουν όλα αυτά τα ζητήματα και θα ήθελα τώρα να σας ευχαριστήσω και έξω όνομα της ομάδας μου και θα δείτε πως η συνεργασία μας θα είναι όντως εξαιρετική αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Νέα Καστήλιο. Κυρία Μπαλούστη, ο Στέρφος Μπαλούστης έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον ε, Υπουργό για την ε, διεξοδική παρουσίαση του προγράμματος της Ιρλανδικής Προεδρίας ε, από την οποία θα αναλάβει η, Προ... Φιλανδία. Γνωρίζουμε ότι μέχρι το 2014 η ιστορική αγορά ενέργειας θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το 2015 ούτε ένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να βρίσκεται απομονωμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη, περίπλοκη, απαιτεί πολλέ επενδύσεις. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά σε ιδιώτε επενδυτέ και ε, υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον αυτέ οι στρατηγικοί στόχοι θα μπορέσουν να επιτευχθούν. Κατά τη διάρκεια της σα, κατά τη διάρκεια τη Λιθουανιακή Προεδρία ε, και ούτω Δεν ε, δεν πολύ για την ενέργεια, για την ψηφιακή ατζέντα, διότι η όλα αυτά τα θέματα έχει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά υπάρχει μια πρακτική διασύνδεση μεταξύ του φυσικού αερίου και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διότι αν δεν έχουμε εναλλακτικά δίκτυα, αυτοί οι πόροι δεν έχουν μόνο οικονομική σημασία, αλλά και πολιτική. διότι αφορούν άμεσα και την ανταγωνιστικότητα και έχω κατά νου τα κράτη της Βαλτικής. Στο πρόγραμμά σας είπατε ότι θα αναπτύξετε δράσεις στον τομέα της ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ή πώς θα μπορούσατε να διευκρινίσετε περαιτέρω πώς θα το πετύχετε. και εφόσον αναγνωρίζετε ότι το σοβαρότερο πρόβλημα σήμερα για την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας ε, είναι ε, η διασύνδεση του φυσικού αερίου με τη δίκτυα ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Ευχαριστώ. Το λόγιο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερα θεαρετικό να ακούμε ότι η Ιρλανδική Προεδρία θέλει να ασχοληθεί με την ε, νέα αγορά και την ψηφιακή ατζέντα. Πάντω οι φήμε που έρχονται από το Συμβούλιο και οι συζήτηση που διαξάγονται στον οίκο μα, μπορούν ε, τελικά να πληγούν ε, τους επόμενους μήνε. Και κινδυνεύει εμπιστοσύνη των πολιτών σε ό,τι αφορά τη δυνατότητά μας να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ιρλανδία πρότεινε ότι αυτή η εμπιστοσύνη εδώ δεν θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις ε, και η οδηγία του 1995 ε, έχει θεωρηθεί ότι ε, παρεμποδίζει την πρόσβαση τους στα, δίκτυα, στα διαδίκτυα. Είναι ενθαρρυντικό το ότι η Ιρλανδική Προεδρία θέλει να εστιάσει στα ευθύ δίκτυα, αλλά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που έχουν υπολοιθεί σε αυτή την Επιτροπή και τις οποίες έχει προωθήσει μια Αμερικανική εταιρεία στον, του κλάδου για τη μέθοδο συλλογή προσωπικών δεδομένων, ενώ γνωρίζουμε ότι έχουμε ευρωπαϊκές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που μπορούν να ε, εφαρμόσουν τα δίκτυα και τους ευθύ μετρητέ. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ακούσουμε περισσότερα σχετικά με τις απόψεις σα περί αυτών των ζητημάτων και το πώ προτίθεστε να εργαστείτε για την βελτίωση τη προστασία δεδομένων για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την εμπιστοσύνη που έχουν επιδείξει μέχρι τώρα οι ψηφοφόροι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίτσεστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καλημερίζω τον κύριο Υπουργό. Χαίρομαι που σας βλέπω. Αργότερα, όπως ακούσατε, θα εξετάσουμε το θέμα της ένισα και τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να επιτευχθεί συμφωνία και φαντάζομαι το Συμβούλιο να δεχθεί τα αιτήματα του Κοινοβουλίου τώρα για το δομέα της ενέργειας. Να πω ότι έχουμε πολλά φιλόδοξα προγράμματα αλλά και γενικότερα φιλοδοξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα αυτό για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ε, να προωθήσουμε την οικονομία ε, χαμηλής εκπομπής ε, του άνθρακα, αλλά όλα αυτά απαιτούν τεράστιες επενδύσεις, ε, οι ευθύς μετρητές, ευθύη δίκτυα, η βελτίωση της πρόσβασης στα φυστάμενα δίκτυα, Ε, δεν θα πρέπει, να πρέπει να σκεφτούμε δε, την αύξηση των επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς. Αλλά γνωρίζουμε πως οι οικονομίες μας αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Πολλές προκλήσεις. Υποστηρίζω τις προτεραιότητες που θέσατε, αλλά πιστεύετε πως έχετε βρει μάλλον τρόπο για να αυξήσουμε την χρηματοδότηση. Ευχαριστώ τον κύριο Τσίτσεστερ. Μετά από αυτή την το πρώτο γύρο παρεμβάσεων από πλευρά πολιτικών ομάδων, το λόγο έχει ο Υπουργό και έπειτα συνεχίσουμε του υπόλοιπου συναδέλφους. Παρακαλώ. Uh, thank ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους σας που έθεσαν κάποιες τόσο σημαντικές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που προσφέρεστε να συνεργαστείτε εκ μέρους της παιδείας για τα θέματα τα οποία σας εξέθεσα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Όλοι σχεδόν αναφέρθηκαν στην εσωτερική ενεργειακή αγορά και την πρόοδο που απαιτείται. Προθεσμία. Όπως ξέρετε, είναι πολύ μικρή. Και κατά εκτίμηση της Επιτροπής πολλές δράσεις ακόμη θα πρέπει να αναλυφθούν. Περισσότερες από 100 δράσεις. 20 αφορούν τις ίδιες τις χώρες μέλη. Υπάρχουν εδώ πολλά θέματα τα οποία αποτελούν πρόκληση, αλλά νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι σε ένα πράγμα. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι είναι απαραίτητο να προοδεύσουμε το συντομότερο δυνατό και όσο περισσότερο μπορούμε ώστε να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά, ακόμη και να αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι πρέπει να σχεδιάσουμε την αγορά με τρόπο που να επιλύει δύσκολα θέματα. Παρά το γεγονός ότι θα πρέπει ίσως τα έργα υποδομής να περιμένουν κάπως περισσότερο. Η κυρία Ντελκαστήλιο ανέφερε κάποιες από αυτές τις προκλήσεις όπως και ο κύριος Τσίτσιστερ στα σχόλια που έκανε. Και βεβαίως ορθά είπε ότι χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις. Δύσκολα όμως μπορεί κανείς σε επίπεδο γετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκεράσει επιχειρήματα που λέγουν επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης, αλλά για να μπορέσουμε να φάσουμε στην υλοποίηση αυτών των στόχων δεν διαθέτουμε τα κατάλληλα κονδύλια, τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωζώνης, η οποία βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. Δεν είναι ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Το πρόβλημα είναι πώς θα τα διοχετεύσουμε στον κατάλληλο τρόπο, ώστε να γίνουν παραγωγικές και επικερδείς επενδύσεις στον τομέα των ενεργειακών. Βεβαίως εδώ Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι έτοιμο να συμμετάσχει ε, και ο ιδιωτικός τομέας σε ενεργειακά θέματα. Όπως είπε και η συναδελφό σας, υπάρχουν χάσματα, υπάρχει έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας και ε, υγραερίου. Και θα ήθελα με εφικτό τρόπο να αντιστραφεί η κατάσταση ώστε να έχουμε κάτι θετικό. Δεν είναι ότι δεν έχουμε λοιπόν τα χρήματα. Στον ε, ενεργειακό τομέα χρειάζεται χρόνος μεταξύ του σχεδιασμού και της εκτέλεσης. Θα πρέπει λοιπόν να παράσχουμε την βεβαιότητα όσο μπορούμε στους επενδυτές για να τους προσελκύσουμε. Εάν υπάρχουν ε, αμφιβολίες όσον αφορά τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής μας και υπάρχει αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών και δεν ξέρουν αν θα αλλάξουμε ρότα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε επενδύσεις. Άρα πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι οι πιο σημαντικές δράσεις τις οποίες μπορεί να λάβει η Επιτροπή και στα πλαίσια αυτών να δημιουργήσουμε την βεβαιότητα. Πρόκειται για μεγάλη πρόκληση και ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Η κυρία Ντεκαστήλιο, καθώς και άλλοι συναδελφοί σας, έστεσαν το θέμα του ΣΕΦ. Το ΣΕΦ βεβαίως, επί αυτού του θέματος, θα συνεισφέρει θετικά τις διευκόλυνσεις δηλαδή για το συνδέοντα στην Ευρώπη δεν ξέρουμε και ούτως άλλως εγώ δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα των συζητήσεων του πολιετούς. Πολύ θα ε, εκπλαγώ αν πρόκειται για βελτίωση τελικά. Εν πάση περιπτώσει, το Φεβρουάριο θα ξέρουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω θα είναι λυπηρό εάν ε, δεν υπάρχει βελτίωση αυτή τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, διότι εδώ έχουμε την ευκαιρία να γίνουν δημόσιε επενδύσει ταυτοχρόνως με ιδιωτικές, ώστε κάποια από αυτά τα κενά τα οποία έχουμε να τα ξεπεράσουμε. Αφού τα εντοπίσουμε πρώτα. Διότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι τα θέματα Εν πάση περιπτώσει, το να δημιουργήσουμε θέσει απασχόλησης, νέε οικονομικέ δραστηριότητες, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε και βεβαίω μέσω πρόθεσμα να μπορέσουμε να έχουμε ε, ενέργεια πιο αποδοτική και για τους ιδιώτες αλλά και για τις επιχειρήσεις. Κάποιοι ομιλητές ανέφεραν και την ένισα. Και συμφωνώ με τον κύριο Τσίσεστερ ότι όντω βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο και νομίζω ότι αργότερα αυτό θα το συζητήσουμε, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η στιγμή είναι πολύ σημαντική. Ή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε ό,τι κάνουμε στα πλαίσια της ΕΝΙΣΑ, διαφορετικά θα θέσουμε ένα αμφιβόλο τον οργανισμό αυτό. Χθε έγιναν συζητήσεις και νομίζω ότι επιτελέστηκε πρόοδος, πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι επιλύθηκαν όλα τα προβλήματα, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε αποδοτικά να δουλέψουμε για να λύσουμε όλα τα εκκρεμή θέματα. Ξέρουμε για ποιο λόγο ο ρόλος της ένισα είναι σημαντικός στον κόσμο των κυβερνοαπειλών και για να εξασφαλίσουμε την ε, ε, ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Η κυρία Anders Ντότερ, που είναι φαν της ε, ποδοσφαιρικής μας ομάδας, στην οποία θα πω ότι μέχρι τότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μέχρι το τέλος της Προεδρίας, αλλά μετά μπορεί να έρθετε ε, ε, σε επαφή μαζί μου. Και ο κύριος ε, Κέλλη, που είναι πρώην πρόεδρος της ομάδας μας, μπορεί να σας βρει εισιτήρια. Καταλαβαίνω αυτά τα οποία λέτε για τα θέματα προστασίας των δεδομένων. Δεν είναι θέμα δικής μου προτεραιότητας και αρμοδιότητας, κυρίως είναι θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου εσωτερικών και δικαιοσύνης. Αλλά γνωρίζω το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του τελευταίου έτους και την σημασία της προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στα πρέσια της ανάπτυξης της, της ε, ενιαίας εσωτερικής αγοράς και της ψηφιακής κοινωνίας. Αν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θέλουμε να έχουν εμπιστοσύνη και να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων και τη ιδιωτική ζωή. Αυτό είναι πρωταρχική σημασία παρά το γεγονό ότι είπα αυτό το θέμα δεν είναι θέμα δική μου αρμοδιότητα. Έχω συζητήσει και θα συζητήσω το θέμα περαιτέρω με τον Υπουργό Δικαιοσύνη που ασχολείται άμεσα με το θέμα αυτό. Μακρηγορώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν ανέφερα κάτι. Ναι. Η ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Ίσως πρόκειται για το πιο σημαντικό θέμα στον αφορά τις τηλεπικοινωνίες σήμερα και θα θέλαμε βεβαίως να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, αλλά δεν θέλω να φανώ ότι είμαι αφελής. Κατανοούμε τις ε, δυσκολίες που υπάρχουν. Εάν μέχρι το μέσον ε, του έτους μπορούσαμε να προχωρήσουμε για να προωθήσουν με τα πράγματα σε επίπεδο ε, Συμβουλίου. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε προβλέψει πολλές συναντήσεις ομάδων και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε θέση του Συμβουλίου. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι πολλές χώρες έχουν διαφορετικές απόψεις, έχουν άλλες συστήματα πιο ε, προηγμένα, άλλες πρέπει να κάνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις. Αλλά πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό φάκελο, τον πιο σημαντικό στα πλαίσια των τηλεπικοινωνιών. Και βεβαίω θα θέλαμε να έχουμε και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί είναι να μπορέσουμε και ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση να διαμορφώσουμε τη θέση του Συμβουλίου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Περάσουμε στον δεύτερο γύρο τώρα των παρεμβάσεων. Ξεκινάμε από τον κύριο Βιντάλ Κουάντρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την εδώ παρουσία σας σήμερα. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία και να σας συγχαρώ για τις θετικές εξελίξεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην Ιρλανδία. Γνωρίζουμε, γνωρίζονται ότι η χώρα έχει πολλούς φίλους στο κοινοβούλιο μας και εσείς αποτελείτε ένα, αποτελέσατε μάλλον ένα μοντέλο σε περίοδο οικονομικής ε, εφορίας και θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή να μας υποδείξετε πώς θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για κάποια από τα νομοθετικά κείμενα που εξετάζουμε και με τα οποία θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια του Ιρλανδικού εξαμήνου. Να σας ευχαριστήσω όμως εφόσον μπορέσετε να μας μιλήσετε για, και να σχολιάσετε γενικά για την ε, ανερχόμενη απογοήτευση των πολιτών μας σε σχέση με ζητήματα ενεργειακής πολιτικής ε. ότι εν ταυτόχρονα Παίζουμε πάρα πολλά όργανα. Έχουμε πολλούς στόχους, πολλές πολιτικές, χρησιμοποιούμε πολλά εργαλεία και ορισμένες φορές ε, αυτή αυτός ο πολλαπλησιασμός των στόχων και ε, νομοθεσίας δημιουργεί σύγχυση. Και εισαγάγει πολύ άχδος γραφειοκρατικό ή οικονομικό στις οικονομίες μας αλλά επίσης μπορεί και να δημιουργήσει ε, ασυναρτησία, θα έλεγα, ανακολουθίες. Λοιπόν, θα μπορούσατε να έχετε μια απλή, απλούστερη προσέγγιση, ορίζοντας έναν κοινό στόχο, π.χ. σε μείωση διοξιδίου του άνθρακα, ή για την φορολόγηση του άνθρακα, των κούμπων άνθρακα. Να υπάρχει ένας κανόνας ε, ίδιος για όλους και όλοι να τον κατανοούν, να υπάρχει και η απαραίτητη ευελιξία για την επίτευξη αυτών των στόχων. Να υπάρχει δηλαδή και μια προσαρμογή ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες ε, και τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Με άλλα λόγια δηλαδή, Υπουργέ δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να προστέψουμε τα πράγματα και να, βάλουμε, να τα βάλουμε σε μία τάξη σε ό,τι αφορά την πολιτική ενέργεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα θέλω να πω δεν είστε εσείς από το δικό μου πολιτικό κόμμα, οι περισσότεροι στην Ιρλανδία θα έλεγαν πάντως ότι ο προεδρεύων είναι από τους πιο έντιμους και ικανούς πολιτικούς. Τα είδαμε και από αυτά που μας είπε σήμερα. Καθώς επίσης και η έπαινη που απίφθινε στην Δανική και Κυπριακή Προεδρία. Τώρα, ανέφερε και ορισμένες σημαντικές εκδηλώσεις, η ΣΕΤ στο Δουβλίνο, που θα γίνουν δηλαδή, είναι επικείμενες, Ο αρμόδιος επίτροπος με έχει προσκαλέσει να έρθω να ομιλήσω για θέματα τα οποία θα είναι σημαντικά για το προς τα που κινούμεθα κτλ. Ο συνάδελφός μου Δεστράτερ έχει φύγει, αλλά ελπίζει να μπορέσει να έχει εισιτήρια για τους τελικούς του χρόνου, για τους τελικούς αγώνες του ποδοσφαίρου δηλαδή. Πάντως, εμείς μιλήσαμε σήμερα το πρωί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την οποία είμαι εισηγητής. Είναι σημαντικό να τονίσουμε και να επαναλάβουμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εξελιχθεί μια κατάσταση όπου θα αναχαιτήσουμε την πρόοδο των ευφυών δικτύων με υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί έτσι ώστε να προκύψει η καινοτομία αυτή και βέβαια η απασχόληση που θα συνεπάγεται. Τώρα, με την ευρύτερη έννοια, το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εξαρτώμεθα υπερβολικά από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Θα ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Υπουργό, τι μπορούμε να κάνουμε στη διάρκεια της Προεδρίας για να εξασφαλίσουμε ποικιλία προμηθευτών και ασφάλεια προμηθειών. και για τις 27 χώρες μέλη. Διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι και διαφορετικές ανάγκες ανά χώρα μέλος. Ευχαριστώ. Κύριε Τοζενόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω κι εγώ κύριε Υπουργέ. Μπράβο σα που τα καταφέρατε και ήρθατε εδώ στην παγωμένη πρωτεύουσα τη Ευρώπη. Δεν είναι και τόσο εύκολο, ούτε μπόρεσαν καν όλοι οι συνάδελφοί μα. Επομένω, εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθειά σα. Είμαι εισηγητή δε για τα α, ε, δίκτυα ευρέω φάσματο υψηλή ταχύτητα. Και θα συναντηθούμε αργότερα, γιατί επιθυμώ πολύ να συζητήσουμε για τι προτεραιότητε για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο θετικό που η χώρα σας, η Ιρλανδία, αναλαμβάνει την Προεδρία της Ένωσης, γιατί έχει μεγάλη εμπειρία με την ανάπτυξη ε, δικτύων ευρέως φάσματος υψηλής ταχύτητας, αλλά και άλλων τεχνολογιών των επικοινωνιών. Γνώση η οποία θα αποδειχθεί πολύ σημαντική όταν θα συζητούμε τα θέματα αυτά. Τώρα έχω μια ερώτηση που είναι κάπως περίπλοκη για το πρόγραμμα SEF, Connection δηλαδή ε, την ε, διευκόλυνση μάλλον ε, συνδέοντας την Ευρώπη. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στο Συμβούλιο σας οδηγούν να βλέπετε με ποιον τρόπο τη μελλοντική εξέλιξη. Θα μπορέσει να βελτιωθεί η διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Αναφέρατε την ανάγκη εξοικονομήσεων και την ανάγκη ανάπτυξης τεχνολογιών επικοινωνιών ακόμη περισσότερο. Πιστεύετε ότι οι χώρες μέλη θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν το πρόγραμμα ή θα παραμείνει περισσότερο στο χαρακτήρα πιλωτικού για το μέλλον. Πώς θα χρησιμοποιηθούν ή πώς θα εξασφαλιστούν οι δημόσιοι πόροι. σε ένα τομέα όπου κυρίως η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η συζήτηση που διεξήχθη ήδη στην Επιτροπή μας ήταν πολύ δύσκολη, πολύ περίπλοκη και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που μπορέσαμε τελικά να συμφωνήσουμε στην ανάγκη να υποστηριχθούν οι βέλτιστες και πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Αναμένω πάντως με μεγάλο ενδιαφέρον τις μελλοντικέ μας συναντήσεις για να συζητήσουμε το θέμα αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. κυρία Ουσμποκ. Ουλσκοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ Ράμπιτ. Συναντηθήκαμε και στο παρελθόν και συζητήσαμε για την σημασία της ταυτοποίησης ε, θέμα με το οποίο, με το οποίο ασχολούμαι και στην Επιτροπή μας. Είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα περίπλοκο. Εμπλέκονται διάφορες επιτροπές σε αυτό το ζήτημα της ταυτοποίησης. Εγώ δεν ε, προβληματίζομαι γι' αυτό. Θεωρώ ότι η συνεργασία μας θα προχωρήσει με τρόπο ομαλό. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ακούσω είναι ποια είναι κατά η θέση που επικρατεί στο Συμβούλιο. Πώς ε, βλέπουν το ζήτημα τα κράτη-μέλη. Ποιες είναι οι δυνατότητες ε, προόδου σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση. Σίγουρα τα βλέπουν τα πράγματα όπως και εμείς ε, γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και περαιτέρω απασχόλησης μια περαιτέρω διασφάλιση για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Φυσικά το συμφέρον είναι κοινό, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική στάση με την ε, εκμετάλλευση αυτού του, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Και μια άλλη ερώτηση που αφορά την ενεργειακή πολιτική. Με χαροποιεί ιδιαίτερα που ακούω ότι εσείς έχετε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα και σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη αναφέρατε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ε, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και παίζει ιδιαίτερο ρόλο όταν πρέπει να αναπτύξουμε νέες αγορές. Οι στόχοι των αγορών θα πρέπει να είναι σαφείς εφόσον θέλουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις σε θέματα ειδικά ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επί του σημείου αυτού είμαι λίγο απεσιόδοξη, διότι δεν κατορθώνουμε να εγκρίνουμε και να υιοθετήσουμε αποφάσεις ε, που να είναι ξεκάθαρες ε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό αντανακλάται και σε άλλους χώρους. Και έχω ερωτήσεις τόσο για το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όσο και για τις ενεργειακές πολιτικές του. Θα κατορθώσουμε να διατηρήσουμε αυτό το τόσο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν αξιόπιστες και βάσιμες ε, προβλέψεις. Η οικονομική κρίση είναι τόσο βαθιά ανά την ώστε χρονοδιαγράμματα όπως ε, αυτά κρίνονται ιδιαίτερα φιλόδοξο. Αλλά όλοι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια έτσι ώστε να πετύχουμε κάτι το απτό. Ίσως θα να μας πείτε κάτι περί αυτό. Ευχαριστώ, ο πρώτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, που βρίσκεστε ανάμεσά μας. Πιστεύω ότι είναι τόσα τα προβλήματα τα οποία είναι και ε, πολύπλευρα. πλευρά χρειάζεται ε, μια, ε, ένα παιχνίδι ομαδικό προκειμένου να δημιουργήσουν συνεργασίες ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Καταρχήν, να σας πω ότι με ενδιαφέρει πολύ το θέμα της προσαρμογής ε, του κλίματος και ε, η προστασία αυτού. Και κατ' εμέ χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε όλο και περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι κατακαιρματισμένες ε, αν την υφήλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί μια ομάδα προσώπων που έχουν συνηθίσει να συνεργάζονται. Τώρα, από πλευράς ε, ανακοίνωσης ε, και, την, για την ασφάλεια των επικοινωνιών, θεωρώ ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. παρατηρούμε πως είναι δυνατόν με αυτές τις επιθέσεις που γίνονται στον κυβερνοχώρο πως μπορούν να ε, επηρεαστούν πάρα πολλά κράτη. Έχω την εντύπωση ότι μπορούν να υπάρξουν και κάποια εξαρτήματα που μπορούν να προσθεθούν στους υπολογιστές αλλά και τηλεπικοινωνίας που δίνουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες και μπορούν να τις ε, μεταφέρουν. Θα ήθελα λοιπόν να με καθησυχάσετε επ' αυτού. Ε, και επίσης ε, να ζητήσω πως τόσο το Συμβούλιο όσο και η Ιρλανδική Προεδρία θα πρέπει να δράσουν προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις για πραγματικά ευρωπαϊκές υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο φυσικά. Αυτό θα ήταν σημαντικό και για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την έξοδο από αυτήν την οικονομική κρίση που μας μαστίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόντι. Ο κύριος Μπουτικόφερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Σα ευχαριστούμε για τι εξηγήσεις σας όσον αφορά τα σχέδια και τι προτεραιότητε τη Προεδρίας σας. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο εσείς δεν αναφέρεται κατά προτερά και δεν νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις προτεραιότητες. Πιστεύω όμως ότι πρόκειται για μια σημαντική συζήτηση για την βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης. Σημαντική συζήτηση. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι όλο και πιο σημαντικό. Το όραμα, ωστόσο, μιας ικανής και ευθύους ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιομηχανία που να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα δεν μου φαίνεται να ολοκληρώνεται. Άκουσα τον Κάμερον σήμερα στην ομιλία του, μίλησε πολύ για ανταγωνιστικότητα, αλλά είχα την εντύπωση ότι αυτός δεν εμπιστεύεται την δύναμη μιας πραγματικής επίθεσης εντό εισαγωγικών για την ανταγωνιστικότητα αλλά ακολουθεί μάλλον άλλο δρόμο. Και το ευρωπαϊκό τοπίο των λόμπι οι, αποφα... οι απόψεις είναι πολύ διαφορετικές. Δεν είναι ενιαίες. Το ίδιο σε ό,τι αφορά την διασύνδεση μεταξύ ευρωπαϊκού εξωτερικού εμπορίου και ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Υπάρχουν πολύ έντονες προστατευτικές τάσεις. Είναι σημαντικό, βρίσκω, για την Ιρλανδική Προεδρία αυτή να μην περιοριστεί μοναχά στις άμεσες επικείμενες προτεραιότητες, αλλά να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να προκαλέσει τέτοια συζήτηση, διότι πρόκειται για μακροπρόθεσμη εξέλιξη. Και ελπίζω αυτή η μακροπρόθεσμη εξέλιξη να μην οδηγηθεί σε εσφαλμένη κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Κυρία Άντρες Μπαρέα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Ε, αναφέρατε ότι κάποιες υποδομές ε, θα πρέπει να περιμένουν και ε, κατά πόσο θα υπάρξουν αρκετά κονδύλια για χρηματοδοτήσεις. Η κυρία Πιλάρ Καστήλιο σας είπε ότι ασχολείται με το ζήτημα και θα ήθελα και εγώ να θέσω το ίδιο ερώτημα. Υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα. Το μέσο δεν, χρησιμο... δεν έχει λόγο ύπαρξη αν δεν υπάρχει κατάλληλη οικονομική στήριξη. Γενικά η κατάσταση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού είναι πτωτική και θα ήθελα να πω το εξή. Τι προγράμματα δράσης προβλέπει η Ιρλανδική Προεδρία και τι στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Τώρα η βιομηχανική πολιτική που παρουσιάστηκε δίνει στην ανταγωνιστικότητα μεγάλη σημασία, αλλά και στην δημιουργία θέσεων απασχόληση. Η απασχόληση που ξέρετε αντιμετωπίζει πολύ σημαντική κρίση. Βρισκόμαστε στην αρχή τη συζήτηση, αλλά θέλαμε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι για την δημιουργία κριτηρίων και για την ενδεχόμενη λύση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει στον βιομηχανικό τομέα η Ευρώπη. Ευχαριστώ, κύριε Μπαρέα. Δεν έχω άλλον εγγεγραμμένο. Να δώσω το λόγο για το τελευταίο κομμάτι της εδώ παρουσίας του στον Υπουργό Ράμπιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις έχουμε. Κύριος Βιδάλ ο πρώτος, σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια για τη χώρα μου. σίγουρα προοδεύσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά δεν θα έλεγα ότι έχουμε εντελώς διαφύγει τον κίνδυνο και θα ήταν μεγάλη βοήθεια αν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, κυρίως με αυτές που έχουμε εμπορικές συναλλαγές υπήρχε οικονομική ανάπτυξη. Και βεβαίως για τις φούσκες πρέπει, στη χώρα μας θα πρέπει να υπομισθούμε την ευθύνη. Όταν κατέρευσε ο οικοδομικός τομέας, ξέρουμε ότι δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα και πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα έσοδα του δημόσιου τομέα. Πολλά μέτρα τα οποία λάβαμε ήταν επώδυνα για τους πολίτες μας και πολλά είπατε κι εσείς για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Ο κυριότερος στόχος είναι η ανάπτυξη και το ανέφεραν και η κυρία Αντρέας Μπαντέα και άλλοι συναδελφοί σας. Όσον αφορά την πρότασή σας, κύριε Βιδαλκουάδρας, αν μπορεί να γίνει απλούστερη η ενεργειακή πολιτική μας. Αχ, Θεέ μου, βεβαίως και θα μπορούσαμε. Και εγώ είμαι πρώτος υποστηρικτής σας επί αυτού του θέματος. Κάποια θέματα όμως δεν μπορούν να γίνουν πιο απλά και η ενεργειακή πολιτική είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Φερρυπίν, πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα ασχολήθηκα με τις αρχές του κανονισμού που πρέπει να γίνουν όσο ε, προχωρούμε προς την ε, ε, πρότυπο των ενεργειακού στόχου το οποίο θέλουμε και στα πλαίσια της ενοποιημένης ενεργειακής αγοράς. Τώρα, κάποια πράγματα μπορεί ίσω να κάνουν τα πράγματα πιο πολύπλοκο από ότι είναι. Τώρα, πιστεύω ότι υπάρχει σαφήνεια και καλύτερη κατανόηση των πολιτικών που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Πρώτα απ' όλα, η δέσμευσή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τι Ανανεώσιμε Πηγέ Ενέργεια, η δέσμευσή μα για ενεργειακή αποδοτικότητα και η ευρεία δέσμευση για την χρησιμοποίηση λιγότερων ε, ε, στερεών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Πολλοί μου θέτουν την ερώτηση και πολύ ευγενικά οι ευρωβουλευτές. Το θέμα της ε, ε θέσπισης στόχων μετά το 2020. Ακόμη δεν έχει ασχοληθεί το θέμα αυτό το Συμβούλιο. Οι στόχοι λειτουργήσαν σωστά και βοήθησαν την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Το 2020 όσον αφορά τις ε, επενδύσεις ε, στην ενέργεια είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστεύουμε. Και εάν μπορούσαμε να αφήσουμε τη θέση μας για το μετά, το 2020, θα είχαμε μία επιστοδρόμηση αν δεν υπήρχε βεβαιότητα. Τώρα έχει αρχίσει η συζήτηση και συνεχίζεται, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και βεβαίως είναι υποχρεωτικό να μπορέσουμε τις δυνατότητες που έχουμε στην Ευρώπη να αναπτύξουμε τις νέες ενεργειακές μας πολιτικές, να έχουμε προγράμματα αποδοτικά στον τομέα της ενέργειας και αυτό συνεπάγεται ότι θα μειωθούν και νέες θέσεις απασχόλησης. Η κυρία Αντρέ Μπαρέα έθεσε ένα θέμα το οποίο επίσης έθεσαν και άλλοι συναδελφοί σας, τη χρηματοδότηση. Ξέρουμε ότι το σημαντικό ε, θέμα εδώ είναι το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Τη στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει σε τέτοια κλίμακα την ε, οικονομική κρίση και αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα, Θα προτιμούσα να μην έχουμε περαιτέρω οικονομικές περικοπές. Αυτό θα προτιμούσα εγώ να γίνει. Και περισσότερα μέσα όπως την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη για να προχωρήσουμε. Αλλά όλα αυτά στα πλαίσια της ενεργειακής αποδοτικότητας θα μπορούσαν να γίνουν με την δημιουργία μέσων, ε, με εταιρική σχέση μεταξύ ιδιωτικού ε, και δημόσιου τομέα, ώστε να μην επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο ο κρατικός προϋπολογισμός, διότι ξέρουμε ότι η υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θέλουν να βαρύνουν περισσότερο τον κρατικό τους προϋπολογισμό και το χρέος τους, αλλά αν μπορέσουν να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, αυτή η οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσε να συγχυστεί επιτυχώς. Και πιστεύω ότι εδώ για τα προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα, δεδομένου ότι πρόκειται και για την ευημερία και καλύτερες συνθήκες ζωή των πολιτών. Uh, Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κέλλη, για την ανάπτυξη των εφιών δικτύων. Και ότι δεν θα πρέπει καινοτόμες λύσεις να μην βοηθούνται από άχθος της γραφειοκρατίας και άλλα προβλήματα. Θέτει το θέμα των εισαγωγών των ε, ορυκτών καυσίμων. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για όλες τις χώρες. Η ασφάλεια της προμήθειας είναι μέρος σημαντικό της ενεργειακής μας πολιτικής. Πάντα υπάρχουν ανησυχίες όταν κανείς εξαρτάται από, εξαγωγέ, εισαγωγές. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα ε, σοβαρό επιχείρημα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πηγών ενέργειας. Και εδώ μπαίνει πολύ σημαντικά και πάλι το θέμα της χρησιμοποίησης των πηγών ενέργειας πολλά μπορούμε να κάνουμε πιστεύω για να μειώσουμε τις εισαγωγές και την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να δουν επίσης τον τομέα αυτό ποιες είναι και οι τάσεις που διαγράφονται παγκοσμίως. και έχει μεγάλες επιπτώσεις στη ΣΥΠΑ και στην διαμόρφωση της ε, τιμής ε, της ενέργειας το θέμα του σχιστόλιθου και της χρησιμοποίησης του. Ξέρετε ότι απαιτούνται κανονισμοί και κανόνες για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σε πηγή ενέργειας τον σχιστόλιθο. δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θέμα που μπορεί να αλλάξει τον γεωπολιτικό χάρτη της, του κόσμου. Και αν γίνουν αυτάρκης, είπα, και ίσως τελικά αρχίσουν να εξάγουν και αυτή την πηγή της ενέργειας, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε και να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, κατά την άποψή μου, στην Ευρώπη. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Τασενόφσκι για πόσο σημαντικά είναι τα ευρυδοζωνικά δίκτυα μεγάλης ταχύτητας. Περιμένουμε την σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής επί του θέματος αυτού. Όπως σας είπα και στην ομιλία μου, στην Ιρλανδία τώρα μόλις αποκτούμε εμπειρία από αυτό το θέμα και έχουμε θεσπίσει εδώ και έξι μήνες μία task force στην οποία συμμετέχουν οι μεγάλες εταιρείε τηλεπικοινωνιών και αξιωματούχοι από το Υπουργείο μου και εγώ και νομίζω ότι ήταν πολύ θετικά αυτά που κάναμε. Μάθαμε πολλά πράγματα για το, από τον τομέα αυτό και η υπεύθυνη του τομέα αυτού από το πώς λειτουργούμε στο Υπουργείο μας. Είδαμε ποια είναι τα προσκόμματα, τα εμπόδια, που δεν μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε τα δίκτυα αυτά ε, ταχαίως και προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Και όσον αφορά την ε, ψηφιακή στρατηγική για το θέμα αυτό, εκ μέρου της Επιτροπής προσδίδεται μεγάλη σημασία και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να προετοιμαστούμε για την πρόσβαση σε αυτό το είδους τα ευρυζωνικά δίκτυα στο μέλλον. Και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε για το πόσο σημαντικό είναι να διατεθούν τα κατάλληλα κονδύλια από τους προπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα οποία λέγονται στη θεωρία να συνοδευτούν από πράξεις με εφικτά μέτρα για την ανάπτυξη. Να λέμε από τη μια ότι θέλουμε ανάπτυξη και από την άλλη να περιορίζουμε τα μέσα τα οποία θα διαθέσουμε δεν είναι σωστό. Το λέω αυτό σχέση αυτά με τα οποία λέξανε εκ μέρους του κυρίου Κάμερον. Και ως Ιρλανδός υπουργό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία να συνεχίσει να βρίσκεται στον πυρήνα της Ένωσης. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι θέμα εσωτερικό για την Μεγάλη Βρετανία. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στρατηγική σημασία η πολιτική μας στον τομέα της βιομηχανίας στην Ευρώπη, διότι είναι το θεμελιώδη σημασία μέσων θα μας επιτρέπει ψη να αντιμετωπίσουμε την μεγάλη οικονομική κρίση που μας στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και η στρατηγική μας σε θέματα βοήθειας των βιομηχανιών θα πρέπει να υποστηριχθεί και να αναθεωρηθεί. Εάν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε και τις συνθήκες απασχόλησης, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όταν έχετε κράτη-μέλη στα οποία το 50% των νέων κάτω από 25 είναι άνεργα, θα πρέπει να το λάβετε υπόψη. Και γενικά η ανεργία μεταξύ των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά υψηλή και θα πρέπει να αποτελέσει το κέντρο του μελήματος όλων μας. Γίνονται. Η κυρία Ολστφαγ ανέφερε και άλλα θέματα που αφορούν την ενέργεια. Ελπίζω και άλλα συμβάντα που θα οργανώσουμε. Ελπίζω ότι θα υπάρχει κοινωνία μεταξύ ημών και ημών για την ειδική ε, συνάντηση, των, ε, την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας που θα γίνει το Μάιο. Και οι συνάδελφοι θα είναι και σε επαφή με το προσωπικό που εργάζεται επίπεδο ένωση για τον κύριο Ραμπόη. Τώρα, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ηλεκτρονική υπογραφή. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ενθουσιασμός εκ μέρους του Συμβουλίου. Οι συζητήσεις που είχαμε ως τώρα σε όλα τα κρατη ήταν απολύτως σαφής όσον αφορά την σημασία της ενίσχυσης και βελτίωσης της εμπιστοσύνης και της ε, εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρχει για αυτό το θέμα. Δεδομένου ότι οι συναλλαγές μέσω ίντερνετ διπλασιάζονται σχεδόν κάθε χρόνο, να μην πω τριπλασιάζονται. Και όλοι γνωρίζουν ότι καταρχάς υπάρχει δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά κάθε χώρα έχει διαφορετικές τις παραδόσεις, κουλτούρα και ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις από κάποιε χώρες για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Άλλε μπορούν, άλλε δεν έχουν. Και μέχρι τώρα στην πρόοδο που έχει επιτεθεί έχουμε δει ότι υπάρχουν θεμελιώδη σημασία θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και διευθετηθούν περαιτέρω. Πρέπει να πω ότι έχουν γίνει ε, προβλέψεις για 10-12 συναντήσεις ομάδων εργασίας για το θέμα αυτό και τα άρχισε πρόεδρε μα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα που να συζητούν. Δεν υπάρχει όμω εκ μέρου των κρατών μέλων έλλειψη πολιτική δέσμευση. Όλοι αναγνωρίζουν πόσο κεντρική σημασία είναι το θέμα αυτό. Και τα θέματα που τέθηκαν σε επίπεδο Συμβουλίου δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά τα οποία έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε δημερώσει συζητήσει μεταξύ μας. Τα θέματα είναι πραγματικά παρεμφερή και θα ήθελα σε αυτό το ειδικό θέμα και σε αυτό το φάκελο να επιτευχθεί όσο μεγαλύτερη πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί. Αλλά πρόκειται για πολύπλοκο θέμα και υπάρχουν δυσκολίες. Κάποια από τα θέματα που έθιξαν πρώτοι και άλλοι. Κοιτάξτε, πρέπει όντως να αρθούν στο επίπεδο του Συμβουλίου οι μεγάλες γραμμές της, της ε, πολιτικής, της δημοσιονομικής πολιτικής και άλλα. Και σίγουρα ο δικός μας Πρωθυπουργό έχει την πρόθεση τα θέματα αυτά να τα θέτει διαρκώς στο Συμβούλιο. Γιατί είναι και τα πιο μεγάλα που αντιμετωπίζουμε. Ξέχασα κανέναν, κυρία Πρόεδρε. Για το θέμα της κυβερνοασφάλειας που απασχολεί πολλούς. Γνωρίζετε ότι η Κομισιόν προτίθεται να δημοσιεύσει έγγραφο στρατηγικής για το όλο θέμα της κυβερνοασφάλειας. Και αυτό θα οδηγήσει εν τέλει σε οδηγία. Θα εξελιχθεί σε οδηγία. Και αυτό τονίζει την ανάγκη να συμφωνήσουμε, αν είναι δυνατόν και όσο γίνεται πιο γρήγορα, στο θέμα του οργανισμού ένισα. γιατί είναι σημαντικός οργανισμός αυτός, εφόσον συζητούμε πρόταση για την κυβερνοασφάλεια, όπως είπα πρέπει να συζητηθεί το θέμα του οργανισμού. Και είπα και πριν ότι θα το συζητούμε με τον κύριο Τσίτσεστερ που σας εκπροσωπεί και εγώ από την πλευρά του Συμβουλίου. Θα το συζητήσουμε μάλιστα σήμερα αργότερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό για τις απαντήσεις που έδωσε στους συναδέλφους. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες ε, να συναντηθούμε. Τώρα, σε ό,τι φορά τις εργασίες μας, γνωρίζετε ότι η συνεδρίασή μας ε, θα, της Επιτροπής θα ξεκινήσει στις 16.00. 3 με 4 έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών οργανώσαμε τη συνέντευξη των συντονιστών μεταξύ 3 και 4, διότι οι υπουργοί που έχουμε προσκαλέσει δεν μπορούν να έρθουν ανάμεσά μας ε, πριν από τις 17.00. Ευχαριστώ, καλή όρεξη. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.